Can we, can we... Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf äh, heute Sie ganz herzlich begrüßen zur gemeinsamen Sitzung. Äh, Ξεκινάμε την κοινή μας ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής ΛΥΜΕ, παρουσία του Επιτρόπου ΣΕΜΕΤΑ. Και το θέμα μας είναι η οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λεγόμενη οδηγία PIF. Είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία. Πρόκειται για μια οδηγία η οποία αφορά πολύ επίκαιρες υποθέσεις αφορά την καταπολέμηση απάτης από την Όλαφ. Σήμερα το πρωί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση για τα θέματα αυτά και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση λειτουργίας της Όλαφ. Η πρόταση λοιπόν της Επιτροπής μέσω αυτής της οδηγίας PIF έχει σκοπό να βελτιωθεί η νομική κατάσταση στην Ευρώπη και να υπάρξει μια καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των, του ποινικού κώδικα των κρατών μελών, μέσω των διατάξεων. Χαίρομαι ιδιαίτερα και χαιρετώ τον Επίτροπο λοιπόν, τον συνεισηγητή Λόπες Αγγιλάρ, που μαζί με την κυρία Γκρέσλε, μέλος της Επιτροπής μας, θα μας παρουσιάσουν το θέμα αυτό. Επίσης χαιρετίζω και τους ε, συναδέλφους από την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και βεβαίως ε, η εκπροσώπηση της Όλαφ είναι κάτι που θα έπρεπε ίσως να μας απασχολήσει, αλλά είμαστε τόσο ε, ευτυχείς που έχουμε τον Επίτροπο που νομίζω ότι θα καλύψουμε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Πρόεδρε Τόιλερ, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι. Ως Πρόεδρος Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ είναι τιμή μου να συμμετάσχω σε αυτήν την ε, διαδικασία με στόχο την εξυπηρέτηση πολύ σοβαρών στόχων που σχετίζονται και με σημαντικό στοιχεία της ποινική νομοθεσίας. Εμείς με την οδηγία αυτή και με την ε, συμβολή του ποινικού ε, δικαίου προστατεύουμε τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό εξηγεί και το μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Και βεβαίως καλωσορίζουμε και την ε, ε, πρόθεση και τον σκοπό της ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού για του Προέδρου του να συμμετάσχει στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο Σέμετα για να κάνει τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αξιότιμα μέλη. Πριν από δύο εβδομάδες το Συμβούλιο ενέκρινε τη γενική προσέγγιση επί της ε, προτάσεως της Επιτροπής του Ιουλίου 2012. Η συνάδελφος Ρέντιν και εγώ ο ίδιος εξηγήσαμε στις δύο επιτροπές σας την ε, ε, αιτιολογία η οποία κρύβεται πίσω από αυτές τις προτάσεις Επιτρέψτε μου τα τρία κεντρικά στοιχεία να τα υπενθυμίσω εδώ. Πρώτος μας στόχος ήταν να καθορίσουμε καλύτερα τα αδικήματα τα οποία αφορούν ε, τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τις συμπεριφορές και λοιπά αδικήματα. Βεβαίως θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να καθοριστούν και ελάχιστες ποινές για τα δικήματα αυτά ε, που θα είναι ε, ε, κυρώσεις οι οποίες θα είναι σωστές, αναλογικές αλλά και αρκούντος αποτρεπτικές. Δεύτερον, οι διαδικασίες ε, να, είναι, ε, να προβλέπουν αρκετό χρόνο και δυνατότητα διασυνοριακής διερεύνησης. Ε, δυστυχώς η γενική προσέγγιση που ενέκρινε πριν από δύο εβδομάδες το Συμβούλιο δεν αντιμετωπίζει τους στόχους μας. Αντιθέτως, στέκεται πολύ πιο χαμηλά από το επίπεδο εναρμόνισης. Τρία είναι τα μελήματά μας όσον αφορά τη γενική προσέγγιση. Πρώτον, το Συμβούλιο θέλει ε, να αφαιρέσει τον ε, ΦΠΑ από το πεδίο εφαρμογής παρότι όλοι οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι ο ΦΠΑ είναι άρκετα συνδεδεμένος με την οικονομική απεικόνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλουμε πραγματικά να προστατέψουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι και η ε, ε, συμπερίληψη όλων των ιδίων πόρων προϋποθέτει και την ε, συμπερίληψη του ΦΠΑ καθώς επίσης και ορισμένα ειδικά εργαλεία δαπανών. Για να είμαστε σαφείς, ο ΦΠΑ δεν μένει έξω από την συνθήκη PIF. Απλώς... The Council not want to introduce και βεβαίως πρέπει να ε, υπάρξουν και ελάχιστες ε, ε, συμφωνίες όσον αφορά de στοιχεία που αναφέρονται σε serious offenses, σε σοβαρά αδικήματα. Κατά αυτήν την έννοια λέμε ότι στη γενική προσέγγιση δεν υπάρχει εναρμόνιση η πρακτική θα σήμαινε ότι στην ουσία, στην πράξη, πολύ λίγα πράγματα θα αλλάξουν ε, και επομένως από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος ή η απειλή φυλάκισης, όλοι θα συνεχίζουν ανενόχλητα να παραβιάζουν τα οικονομικά συμφέροντα. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν ε, και ε, κάποιες, ε, κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι θα είναι συμβατικοί περιορισμοί. Αυτοί όμως δεν θα βοηθήσουν πολύ στην πράξη. Επιτρέψτε μου στο τέλος να πω και ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά την νομική βάση. Το προηγούμενο ε, φθινόπωρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επέλεξε ως νομική βάση το 325 παράγραφος 4 των συνθήκων. Εκεί ακριβώς αναφέρεται ε, η ειδική πρόνοια της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων βάσει επιβολής ποινών που θα είναι δίκες, αναλογικές αλλά και αποτρεπτικές. Γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο απέρριψε αυτήν την νομική βάση ε, υπέρ του άρθρου 83 παράγραφος 2. Η συζήτηση δεν είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα μονάχα. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ο ε, ενωσιακός προϋπολογισμός ε, θα εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κράτη-μέλη. Η Ιρλανδία και η Δανία επίσης αποκλείονται από την δικαστική συνεργασία. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από εμά. Πρέπει να προστατέψουμε ε, τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της ε, και ε, πρέπει η προστασία να είναι σωστή και αποτρεπτική. Αυτό το καταστήσαμε σαφές ε, στην συνάντηση με το Συμβούλιο. Τώρα θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει μια ε, σαφή, ε, σταθερή θέση όσον αφορά το θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά συμμετέχει πλήρως στην διεργασία για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που έχει έτσι ώστε να φτάσουμε σε πλήρη εναρμόνιση στον τομέα που μας απασχολεί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος, ε, για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Τώρα θα δώσω το λόγο στους εισηγητές. Ε, θα δώσω, ε, θα ήθελα μάλλον να δώσω και τον λόγο στον αρμόδιο εισηγητή της Επιτροπής Γιούρι, αλλά νομίζω πως δεν είναι εδώ ακόμα. Αρχίσουμε με την εισηγήτρια από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, την κυρία Γκέρσλε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ επιμείναμε να έρθετε γιατί θεωρούμε ότι αυτή η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου είναι πραγματικά κάτι που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο σε αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακούσαμε, ιδιαίτερα για τη νομική 3254 και όχι 382. Είναι πολύ συγκεκριμένε οι δυνατότητε που έχουμε επιλέγοντας αυτήν την νομική βάση και θα ήθελα επίσης να πω ότι σκοπός μας είναι να καταπολεμήσουμε αυτές τις απάτες και κάθε φορά να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για υποθέσεις οικονομικές, για πρόστιμα, για κυρώσεις που αφορούν άμεσα τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ήμασταν κατά της αλλαγής της νομικής βάσης. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε στην επιλογή μας και να έχουμε κοινή θέση, να δημιουργήσουμε ένα ωραίο αλλά και σταθερό νομικό πλαίσιο το οποίο να μπορούμε να υποστηρίξουμε και Επαναλαμβάνω ότι το 325/4 είναι μια νομική βάση στην οποία θα επιμείνουμε. Εμείς σαν αρμόδια αρχή νομοθετική, σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα επιμείνουμε σε αυτό και κάθε φορά που υπάρχουν προσπάθειες από το Συμβούλιο να αλλάξει αυτό, εμείς θα εκφράσουμε την αντίστασή μας, την αντίρρησή μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα και αυτή η δυνατότητα opting out παρέκκλησης δεν θα πρέπει να δοθεί σε κανένα κράτος μέλος, διότι η νομική βάση 380 παράγραφος 2 περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες και ουσιαστικά θα αποδυναμωθεί πάρα πολύ η διαπραγματευτική μας θέση αν επιλέξουμε κάτι τέτοιο. Θα περιοθεωριοποιηθούμε και αν υπάρχουν τελικά, συνυπάρχουν δύο νομικές βάσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί παρά να έχει περαιτέρω αρνητικά αποτελέσματα. Έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου της 25ης Φεβρουαρίου του 2013 που πραγματικά ενισχύει αυτή μας τη θέση. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να κάνω μια έκκληση προς όλους τους συναδέλφους. Μου φαίνεται πραγματικά ότι είναι πολύ σημαντικό να συσπηρωθούμε εδώ γύρω από αυτή τη θέση. όσο δεν έχουμε βεβαίως ε, ψηφίσει στην Ολομέλεια, για μένα όλα παραμένουν ανοιχτά. Είναι καθοριστικό το θέμα αυτό. Και το συζητήσαμε αυτό και στην πολιτική μας ομάδα. Επαναλαμβάνω, το Συμβούλιο για άλλη μια φορά έδειξε ποιες είναι οι προθέσεις του. Η πρόληψη της απάτης στο άρθρο 1, 2, 4 προσπαθεί να ενσωματώσει όλες αυτές τις ε, δραστηριότητες, διαφθορά, ενεργός διαφορά, παθητική διαφθορά, νομιμοποίηση παράνομων κονδυλίων, κονδυλίων προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε εδώ την θέση μας η θέση της Επιτροπής περιέχει πολύ ουσιαστικά σημεία και μπορούμε απλώς να τη βελτιώσουμε. Άρθρο 2. Το έχουμε συζητήσει. Επαναλαμβάνω το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας λέει εδώ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιοριστούμε μόνο στον προϋπολογισμό να συμπεριλάβουμε όλες τις δραστηριότητες στην οποία είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας Ευρωπαϊκών Επενδύσεων, Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας και άλλων φορέων. Υπάρχουν κάποιες πτυχές ακόμα με σχετική νομική ασάφεια, αβεβαιότητα. Νομίζω όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει όπως το άρθρο 4 όσον αφορά την μετάδοση πληροφοριών να υπησέλθουμε σε θολά νερά, από νομικής απόψεως ε, εννοώ θολά νερά, σε ασάφεια. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε αυτά τα σημεία, άρθρο 4. Επίσης, θα πρέπει να προσπαθήσουμε εδώ να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ του κοινοτικού δικαίου και της νομοθεσίας των κρατών μελών. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει, θα ήθελα να έχω περισσότερες ε, πληροφορίες, ιδιαίτερα όσον αφορά την υλοποίηση όλων αυτών ε, στα κράτη-μέλη, αν υπάρχουν διαφορές, αν υπάρχουν ε, στοιχεία, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στοιχεία για το τι συμβαίνει από εκεί και πέρα στα κράτη-μέλη, αν ε, υπάρχουν κράτη-μέλη παραδείγματος χάρη, τα οποία θα πρέπει να διοθετήσουν συμπληρωματικά ή περαιτέρω μέτρα για την εφαρμογή και την υλοποίηση όλων αυτών και τη μεταφορά τους στην νομοθεσία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να απαιτήσει να υιοθετηθούν αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Υπάρχει αν θέλετε εδώ μια νομική τάξη σε δύο επίπεδα, ευρωπαϊκό, εθνικό. Αυτή η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου, αν θέλετε, είναι κάτι που θα πρέπει να προχωρήσει ακόμα ένα βήμα και αυτό βεβαίως στην πράξη πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες επιπτώσεις. Επαναλαμβάνω, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε αν υπάρχουν ακόμα σημαντικές διαφορές από το ένα κράτος στο άλλο. Θα ήμουν ευγνώμων αν ο Επίτροπος μας έδινε κάποια στοιχεία γιατί είμαι σίγουρη ότι η Επιτροπή τα έχει ήδη επεξεργαστεί όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκρέσλε, την εισηγήτριά μας. Και τώρα ο εισηγητής από την Επιτροπή Λίμπε έχει το λόγο. Thank you, Chairman I would like you... I would like to... Σε ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος θέλω να απευθύνω συγκεκριμένα ερωτήματα στον Επιτρόπο μέτα. Πρώτα απ' όλα, ένα ερώτημα σχετικά με την Όλαφ. Όταν είχα μετάσχει στις συναντήσεις ε, των σκιωδών ε, σχετών και του εισηγητή για αυτό το θέμα, ε, το είχα θέσει και θα ήθελα να ξέρω πόσο αποτελεσματική είναι η σχέση μεταξύ των διοικητικών διαδικασιών της Όλαφ και της ε, Αγγελία ε, Ποινικών ε, Κυρώσεων. από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές των κρατών μελών. Τι ποσά δηλαδή θέλει η Όλαφ να επιστραφούν μετά από την όλη αυτή διαδικασία και τι αντιστοιχεία υπάρχει με τις ποινικές κυρώσεις. Σε ό,τι αφορά την νομική βάση, Βέβαια, εδώ δεν είμαστε για να ξανασυζητήσουμε τα, τη νομική βάση. Θα ήθελα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας μιλήσει λίγο για την ευελιξία και την ετοιμότητα να συμφιλειωθούν τα νομικά επιχειρήματα που ξεκίνησαν ε, να ακούγονται όταν ε, έθεσε το Συμβούλιο το 83. Οπότε ενδεχομένω θα υπήρχε η εξαίρεση κάποιων κρατών μελών, από την out. Και τέλος, θα ήθελα να μου πείτε ως προς τον ορισμό των οικονομικών συμφέροντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πλήρης, είναι διεξοδικό σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Και τις πηγές χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. There is an argument there too. Σε ό,τι αφορά και το φόρο προσθέμενης αξίας. Έχουμε μία πρόταση προεξάρχουσα από την Κομισιόν που όμως το Συμβούλιο δεν δείχνει να θέλει να συμπεριλάβει στη δική του προσέγγιση για το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει η Κομισιόν πώς αντιλαμβάνεται το όλο ζήτημα του φόρου θέμης αξίας. Τι πλονεκτήματα ή τι μειονεκτήματα θα είχε η συμπερίληψή του στην πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είδα τον κύριο Σφίσκα. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Όχι. Τότε θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο, ο οποίος μπορεί να απαντήσει σε αυτά που άκουσε από τους ε, εισηγητές μας. Um, well, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκρέσλε για την υποστήριξη που εκφράσατε στην πρότασή μας. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη ότι είναι μια κρίσιμη πρόταση ότι αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι και ο λόγος ακριβώς για τον οποίο είμαστε και τόσο φιλόδοξοι. Και δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ε, επακόλουθη νομοθετική διαδικασία. Με τα χαράς να σας ε, παρουσιάσω τις συμπληρωματικές πληροφορίες, να σας τις υποβάλω. Ουσιαστικά όλες αυτές τις πληροφορίες στις οποίες αναφερθήκατε τις αναλύσαμε στο πλαίσιο της μελέτης αντικτύπου, που είναι διαθέσιμη, αλλά ίσως θα ήταν χρήσιμο να σας παρουσιάσουν ε, οι εμπειρογνώμονές μας τα κύρια πορίσματα της ε, μελέτης αντικτύπου και τις διαφορές μεταχείρισης και χειρισμού των διαφόρων αξιόπινων πράξεων από τα κράτη-μέλη. Σε κάποιες δεν υπάρχουν χώρες, δεν υπάρχουν ελάχιστες ποινές, ποινικά δικαιώματα που σχετίζονται με την προστασία των οικονομικών συμφέροντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε άλλες χώρες υπάρχουν μόνο διοικητικές ε, κυρώσεις, ποινές χαμηλές ως προς ε, το χρηματικό ποσό. Γι' αυτό και επιτρέπεται πολλές φορές ε, ε, κατά κάποιο τρόπο μια διασυνοριακή επιλογή της καλύτερης δυνατής ε, λύσης για τη χαμηλότερη ποινή από ορισμένους. Εγώ αυτό το οποίο προτείνω είναι να διοργανωθεί ένα εργαστήριο όπου οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα σας παρουσιάσουν αναλυτικά τα πορίσματα της μελέτης αντικτύπου στους συζητητές, τους και όσους συζητητές έτσι ώστε να ενημερωθείτε και να καταλάβετε σε μεγαλύτερο βάθος τα πορίσματα της μελέτης αντικτύπου. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ερωτήματα πόσο αποτελεσματικές είναι οι δράσεις σε επίπεδο κρατών μελών, σε συνέχεια των ε, ερευνών της Όλαφ ε, και τις εθνικές ποινικές διαδικασίες κτλ. Εδώ μπορώ να σας αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Το έχουμε συμπεριλάβει και στη μελέτη αντικτύπου έχουμε 19% follow-up στην περίπτωση της Ελλάδας για παράδειγμα και 91% follow-up στην περίπτωση της Φινλανδίας. Βλέπετε λοιπόν ε, τις πολύ μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά το follow-up. Και αυτό είναι Και αυτό εξάλλου γιατί Ακόμη δεν έχουμε ένα ποινικό δίκαιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είχαμε, θα μπορούσε να εφαρμοστεί μετά από τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την νομική βάση και τα επιχειρήματα σχετικά με την νομική βάση. Δεν είμαι δικηγόρο βέβαια, αλλά νομίζω η νομική υπηρεσία της Κομισιόν έχει υποστηρίξει με πολύ έτσι, εμπεριστατωμένο τρόπο γιατί εμείς επιλέγουμε το άρθρο 325 εδάφιο 4 ως δομική βάση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψη μεταξύ άλλων ότι η προηγούμενη βερσιόν ε, της συνθήκης, συνθήκη της Νίκαιας, απέκλειε ρητός ε, τα ποινικά δικήματα από το άρθρο 280 που αντικαταστάθηκε από το 325. Επομένως, αυτό σημαίνει και έτσι ερμηνεύσαμε και εμείς τα πράγματα ότι θεωρήθηκε με τις συνθήκες Λισαβόνας ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων και κατά το ποινικό δίκαιο πλέον πρέπει να ε, διέπεται από το άρθρο 325 δάφιο 4 της συνθήκης. Το δεύτερο επιχείρημα, το οποίο νομίζω ανέφερε και η κυρία Γκρέσλε, είναι ότι έχουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Με το άρθρο 83, εδάφιο 2 νομική βάση, καταλήγουμε σε διαφορετική αντιμετώπιση του ίδιου αδικήματος σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Δύο κράτη-μέλη και συγκεκριμένα Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία έχουν opt-in αυτή τη δυνατότητα. Η δε Δανία έχει δυνατότητα opt-out από τη διάταξη αυτή, εξαίρεσης. Άρα αυτές οι χώρες θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται μόνο από τη σύμβαση PIF και όχι από την οδηγία. πετεθεί σε ισχύ και αν τελικά βέβαια το 83-2 είναι το άνθρωπο που θα έχει επιλεγεί ως νομική βάση. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ομοιογένεια, την ισότιμη μεταχείριση των ποινικών αδικημάτων. Όταν μιλάμε για το ίδιο ακριβώς έγκλημα, την ίδια αξιόπινη πράξη, που πρέπει να αντιμετωπίζεται εξίσου σε όλα τα κράτη-μέλη. Και το 325.4 ακριβώς αναφέρεται στα κράτη-μέλη, στο σύνολό τους, σε όλα τα κράτη-μέλη. Και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτό το επιχείρημα για το άρθρο 325 ως νομική βάση. Ως νομική βάση για την πολύ σημαντική αυτή νομική πρόταση. Έπειτα έχουμε το ζήτημα των εσόδων. Και συγκεκριμένα το ζήτημα του ΦΠΑ θα γνωρίζετε ότι είμαι αρμόδιος όχι μόνο για την καταπολέμηση της απάτης, αλλά και για τη φορολογία. Πρέπει να σας πω ότι ακριβώς επειδή έχουμε τον ΦΠΑ ως ίδιο πόρο του προπολογισμού της Ένωσης, ακριβώς για αυτό το λόγο ασχοληθήκαμε με πολλέ παραβάσει ε, στα κράτη-μέλη, ακριβώ για αυτό το λόγο όπω είπα, επειδή είναι ίδιο πόρος της Ένωσης ο ΦΠΑ. Και πολλές φορές από τις αποφάσεις του δικαστηρίου αναγνωρίζεται και γίνεται ειδική αναφορά στο ΦΠΑ ως ίδιο πόρο. Και αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την αρμόνιση ορισμένων πρακτικών στον τομέα του ΦΠΑ. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο ΦΠΑ πρέπει να εντάσσεται σε αυτήν την οδηγία. Καλούμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει τη θέση της Κομισιόν. Yeah, thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ποιος θα ήθελε να θέσει ερώτηση ή να κάνει κάποια σχόλια. Δύο. Ο κύριος Ντε και ο Ζων Πιέγοντι έχουν ζητήσει το λόγο μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ βεβαίως και τον Επίτροπο. Σήμερα το πρωί στην ε, Επιτροπή μας είχαμε μία ακρόαση με το Γενικό Διευθυντή της Όλαφ όπου αναφέρθηκαν πολλές ανησυχίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η Όλαφ μια συγκεκριμένη υπόθεση. Το όλο ζήτημα βασίζεται το στατιστικό στοιχείο ότι από ό,τι φαίνεται 43% των εκθέσεων της Όλαφ δεν ε, την χάνουν καμία συνέχεια. Το συζητήσαμε αυτό και με το Γενικό Διευθυντή, γιατί μας φαίνεται πολύ σημαντικό στοιχείο. Πέραν τούτου, δεν είναι σωστό να πούμε ότι 43% δεν είχαν follow-up. Θα πρέπει να δούμε και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Νομίζω ότι και στην αξιολόγηση επιπτώσεων προσπαθήσατε να δείτε τι γίνεται στα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά δεν είδα να κάνετε κάτι για τη λειτουργία της Όλαφ. Σήμερα το πρωί λοιπόν ρώτησα ως μέλος Επιτροπής ε, Κοντ είπα το εξή. Μπορούμε να έχουμε μία εξωτερική μελέτη για την λειτουργία της Όλαφ ε, σε μεμονωμένε περιπτώσεις ε, στα κράτη-μέλη, κυρίως μία μελέτη ποιότητος, δηλαδή που θα αφορά την ποιότητα των ετοιμάτων. Τελικά ε, η μομφή θα πρέπει να αφορά τα κράτη-μέλη αποκλειστικά ή μήπως και στην περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που εξετάσαμε σήμερα το πρωί, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι και η Όλαφ δεν είναι πολύ καλή και ότι ο Γενικό Αγγελέα και οι ιδιοκτικές αρχές ε, των κρατών μελών δεν μπορούν να κάνουν κάτι γιατί έχει υπάρξει και παραβίαση των δικαιωμάτων των ε, υποέλεγχο ατόμων. Βεβαίως εδώ έχουμε ένα ζήτημα με την ε, νομική βάση, αλλά όπως και η Επίτροπος Ρέντινγκ είπε σε μια συνεδρίαση ΛΥΜΠΕ, εάν ε, υποβάλλεται, ε, μάλλον εάν αναφέρεται εδώ ελάχιστες ποινές και μάλιστα είπατε κι εσείς ο ίδιος ότι υπάρχει διαφοροποίηση ποινών και μόνο σε λίγες χώρες υπάρχει αυτή η έννοια των ελαχίστων ποινών. Εμείς θα θέλαμε ε, μία πρόταση της ε, Κομισιόν οριζόντιας ε, διάστασης. Ενώ λοιπόν θεωρούσαμε ότι θα κάνετε μία πρόταση για γενικότερη τροποποίηση του νομικού πλαισίου στις διάφορες χώρες, τελικά βρισκόμαστε με μία ελάχιστη ποινή τότε θα πρέπει να κάνουμε και ελάχιστη ποινή για φόνο και για ανθρωποκτονία και για άλλου είδους ε, αδικήματα. Επίσης, ε, Επομένως, να συνοψίσω, ε, βλέπετε την πλευρά των κρατών μελών, δέστε λίγο γιατί γίνεται και την άλλη πλευρά. Και δεύτερον, αυτό το ζήτημα με τις ελάχιστες ποινές θα το συνεχίσετε. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Ο συνάδελφος Ζωάν Πιεροντή να πάρει το λόγο τώρα. Ο Ζωάν Πιεροντή λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο σύστημα, ε, θέμα, συγγνώμη, το οποίο άπτεται και του ε, ποινικού δικαίου ε, και που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Μια ερώτηση προς τον κύριο Επίτροπο εδώ μας απασχολούν οι απάτες και οι παράνομες δραστηριότητες ή αποκλειστικά ε, οι απάτες. Γιατί στο άρθρο 325 παράγραφος 4 ε, αναφερόμαστε στις ε, απάτες αλλά και γενικότερα σε παράνομες δραστηριότητες ενώ στην οδηγία ε, γίνεται αναφορά μονάχα στις απάτες. Κάνετε κάποιο διαχωρισμό ή μήπως οι παράνομες δραστηριότητες εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας. Δεύτερο, δεύτερη ανησυχία μου δεν έχει υπάρξει διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, βλέπω ότι έχετε έρθει σε επαφή με τους ε, εμπειρογνώμονες, τα εθνικά κοινοβούλια κτλ. Ε, συγγνώμη, ένα σωρό εμπειρογνώμονε ε, και, και εκπροσώπους ε, των φορολογουμένων, αλλά δεν βλέπω να έχετε έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όσον αφορά τον ΦΠΑ, δεν νομίζω ότι είναι ίδιος πόρος ο ΦΠΑ. Έχουμε πει ότι ήδη οι πόροι είναι οι δασμοί ο ΦΠΑ βεβαίως αποτελεί ένα έσοδο για την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, αλλά πέραν τούτου θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο την ομολογία και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δεν την γνωρίζω. Όσον αφορά το άρθρο 12 και την παραγραφή, νομίζω ο, ότι και όσον αφορά και τις ε, προδιαγραφές. Ε, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση. Το έλεγα και πολύ παλιότερα σε μια επιστολή στον Πρόεδρο Μπαρόζο. Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση και όσον αφορά το αστικό και όσον αφορά το ποινικό δίκαιο. διότι οι προδιαγραφές ε, και οι προϋποθέσεις ε, είναι εντελώς διαφορετικές με αποτέλεσμα να χάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ε, επομένως, εναρμόνιση εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Οντή είπε δύο πολύ σημαντικά πράγματα και τα στηρίζω τα υποστηρίζω. Θα ήθελα να λάβω υπόψη μου και αυτό που είπε ο Επίτροπος όσον αφορά τη συνεργασία με το Συμβούλιο που είναι απαραίτητη. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει εδώ να συμπεριλάβουμε και την ε, συνεισφορά των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για όλα όσα κάνατε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και θεωρώ ότι είναι θεμητό ε, να υπάρξει εναρμόνιση της ε, νομοθεσίας ε, και του ποινικού δικαίου όσον αφορά τις καταχρήσεις και παραβάσεις οι οποίες αποβαίνουν προς ζημία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω ότι στη χώρα μου στην Πολωνία, αλλά ίσως και όχι μόνο στην Πολωνία, τώρα τελευταία έχουν υπάρξει ετοιμιγορίες ενδιαφέρουσες του δικαστηρίου οι οποίες ε, αναφέρουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει φορολογική δίωξη ε, ακόμα και για τον ΦΠΑ εάν δεν έχει προηγουμένως αποδειχθεί η απάτη. Και από την ε, Πολωνία λοιπόν για το θέμα αυτό φτάνουν πάρα πολλές πάρα πολλά παράπονα. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ε, ε, πρέπει να πληρώσουν ε, κυρώσεις και χρήματα τα οποία αφορούν απάτες ή παραβιάσεις, χωρίς όμως να έχουν τελεσιδικήσει οι αποφάσεις στα δικαστήρια και να σας πω ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών είναι τέτοιος που πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις κοινέ. Οποιοςδήποτε δεν κάνει ε, ηθελημένα απάτη, οποιοςδήποτε δεν διαπράττει τέτοιου είδους αδικήματα ε, δεν θα πρέπει πριν τελεσιδικήσει η περίπτωσή του και αποδειχθεί η ε, απάτη την οποία τον κατηγορούν, δεν θα πρέπει, λέω, να υφίσταται οποιαδήποτε τιμωρία και κυρίως δεν θα χρειάζεται, δεν θα πρέπει να καταβάλει τα πρόστιμα. Ο κύριος Βαλσίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα και ιδιαίτερα περίπλοκο. Κανείς δεν ζητάει από τα κράτη-μέλη να τροποποιήσουν το ποινικό τους ε, δίκαιο. Όταν ε, γίναμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς τροποποιήσαμε ε, με πολύ θετικό τρόπο το νομικό μας σύστημα. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε η ζωή μας και μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχει απλά η πολιτική βούληση έτσι ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Σε ορισμένες χώρες μέλη για κάποιες παραβάσεις ή αδικήματα δεν προβλέπεται καμία κύρωση ή προβλέπεται απλώς κάποιο χρηματικό πρόστιμο και τελείωσε το ζήτημα. Νομίζω λοιπόν ότι τούτη η πρόταση είναι μια πρόταση που έρχεται τη σωστή στιγμή και πιστεύω ότι στόχο έχει την εισαγωγή ενός συστήματος που ε, θα, εφαρμόζει τουλάχιστον ελάχιστες ποινές όταν ε, υπάρχει απάτη. Στα πλαίσια της ΠΥΦ τώρα τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να δώσουν πληροφορίες οι οποίες να αφορούν περιπτώσεις απάτης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εκθέσεις για τα θέματα αυτά, δηλαδή για την έλλειψη ε, πληροφόρησης ε, που ε, μας εμποδίζει να ταυτοποιήσουμε τον πραγματικό όγκο των απατών. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή την ιδέα των ελαχίστων ε, ποινών σε όλες τις χώρες. Ευχαριστώ κύριος Μιούλντερ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Δεν ξέρω αν κατάλαβα ε, ή δεν το άκουσα τέλο πάντων. Άκουσα... Γίνεται λόγος για ένα είδος ευρωπαϊκού όταν λέμε για τα οικονομικά συμφέροντα, αυτό ε, είναι συνθήκη. Αυτό το ρόλο ε, τον έχει αυτό το άτομο και δεν ξέρω μήπως δεν κατάλαβα. Δεν ε, είδα κάποιος να εκφράζεται πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο, η συγγήτρια, η κυρία Γκρέσλερ. Κοιτάξτε, κάνω μια ερώτηση στον συν εισηγητή. Γιατί η Επιτροπή ΛΥΜΕ ακολουθεί εδώ το Συμβούλιο και είναι υπέρ της αλλαγής της νομικής βάσης. Γιατί δεν ε, συμφωνείτε με την αρχική μας ε, θέση και δεν στηρίζετε την ε, θέση που πρεσβεύει η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Πρόεδρος, θέλετε να απαντήσετε αμέσως. έχουμε ξαναπεί ε, πάνω από μια φορές. Και με εκπλήσει που επιμένετε να μου υποβάλλετε συνέχεια το ίδιο ερώτημα. Την πάτε την έχετε ακούσει επανειλημμένος. Πρώτα απ' όλα είναι γνωμοδότης της Γιούρη. Η Επιτροπή Γιούρη είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή για να αποφασίσει εκ μέρους του Κοινοβουλίου για την νομική βάση. Η Γιούρη έχει την τελευταία λέξη. για την ε, κατανομή των αρμοδιοτήτων. Και δεν είναι ούτε αυθαίρετες ούτε παράλογες ε, οι αποφάσεις. Σίγουρα έχουμε το ποινικό δίκαιο που αυτό εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. up Ορισμός λοιπόν των αξιόπινων πράξεων, επιβολή ε, κυρώσεων. Αυτό είναι μέσα στο ποινικό δίκαιο, αλλά δεν άκουσα κάτι για τη νομική βάση εδώ. Ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει διαφωνία. Εμείς γιατί ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε ακριβώς για να ακούσουμε τις απαντήσεις του Επιτρόπου σε μέτα. Δεν ήρθαμε για να ξανα αναστήσουμε αυτό το θέμα, αυτό το ζήτημα της νομικής βάσης. Συνεργαζόμαστε, πηγαίνουμε χέρι-χέρι δύο επιτροπές. Πρόεδρος, να Επισημάνω κάτι που μόλις ανέφερε ο συνάδελφος Λόπεθ Αγγίλαρ. Έχουμε καταλήξει σε μια κοινή βάση εργασίας μεταξύ των δύο επιτροπών, Λίμπε και Κοντ. Σας παραπέμπω στις ε, συζητήσεις ε, των πέντε των επιτροπών. Εκεί θα δείτε ότι η Γιούρη είχε ζητήσει και είχε πει ότι αυτή έχει την ε, αρμοδιότητα, όπως είπε και ο πρόεδρος Λόπεθα Γίλαρα, και θεωρούσε ότι το 83 εδάφιο 2 πρέπει να είναι νομική βάση. Τώρα ακούμε από τον Επίτροπο Σεμέτα, σε αυτή την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Λιμπεκιακών, ότι η Κομισιόν το σκέφτηκε εντελεχώς και θεωρεί το 325-4 είναι κατάλληλη νομική βάση. Εγώ θα ήθελα να προτείνω. Αν στην διαδικασία ε, συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, μπορούμε να το ξαναθέσουμε. Εμεί είχαμε τι απόψει μα στη, ε, στη διάσκεψη των Αμπρών των Επιτροπών. Δεν πέρασε η απόψή μα, το αποδεχθήκαμε. Τώρα το θέμα οργανωτικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντως ε, πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Η απόφαση πρέπει και θα ληφθεί στην Ολομέλη. Αλλά νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, συζήτησή μας και στην ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο. Αυτό έχω να πω ε, προκειμένου. Πρόεδρο Ελόπε Αγγιλάρ. Ναι, συμφωνώ. Απλά έχουμε μια κατάσταση που πρέπει να την ε, ξεκαθαρίσουμε. Δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ακόμη. Επαναλαμβάνω, γιατί ήρθαμε εδώ. Ακριβώ συμφωνώ. Ήρθαμε για να ακούσουμε τον Επίτροπο. Και γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή διάλεξε το 325 ως ε, την κατάλληλη νομική βάση. Η Επίτροπος Ρέντινγκ ε, εξήγησε το λόγο όταν παρουσίασε την πρόταση Η Επιτροπή Λίμπε. Είχε μπει για το άρθρο 325. Μετά η Επιτροπή Γιούρι γνωμοδότησε κάπως διαφορετικά και αυτό έφερε την αλλαγή. Ε, στη... Σίγουρα είμαστε ε, συνεργάσιμοι και ανοιχτοί. Και μπορούμε να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε το θέμα της νομικής βάσης πρώτη. μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε. Κυρία Γκρέσι, έχετε το λόγο. Συνάδελφε, νομίζω ότι εγώ μπορώ να δεχτώ αυτό που λέτε, πολύ περισσότερο από αυτό που λέτε εσείς, ε, σχέση με την δική μας πρόταση. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση στην Ολομέλεια. Ξέρουμε ποια είναι η γνώμη της ε, Γιούρη. Το θέμα λοιπόν είναι ανοιχτό και αν υπάρχει δημοκρατική, αν θέλετε, λειτουργία αυτού του οργάνου, τελικά η απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια. Γιατί λοιπόν εδώ ζητάτε να φημωθεί το Κοινοβούλιο. Και επιτρέψτε μου, αφού είναι εδώ η Επιτροπή, να το αναφέρω. Και το αναφέρω γιατί πραγματικά θεωρώ ότι μια καλή συνεργασία, μια καλή κοινή λύση είναι πολύ καλύτερη από την εξουρανού λύση. Συμφωνώ, συμφωνώ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Πρόεδρος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το θέμα της φήμωσης είναι θέμα που αφορά την Επιτροπή Άγκρη. Ναι, είναι κάτι που αφορά τα ζώα. και θα πρέπει σαφώς να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα. Το θέμα θα συνεχίσει να συζητάτε εδώ στο Κοινοβούλιο. Οι τρεις επιτροπές είναι ελεύθερες να γνωμοδοτήσουν και στην Ολομέλεια θα ληφθεί η τελική απόφαση. Ο Επίτροπος έχει το λόγο για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και σε όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις, αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το σημείο αυτό. Θα προσπαθήσω λοιπόν πολύ σύντομα να απαντήσω όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της όλα, όσον αφορά την παρακολούθηση και τη συνέχεια που δίδεται στις εκθέσεις. Η μελέτη αντικτύπου γίνεται από εξωτερικούς φορείς και αυτοί οι εξωτερικοί φορείς έχουν αξιολογήσει τα προβλήματα που προκύπτουν στις διάφορες έρευνες της Όλαφ, για ποιους λόγους αυτή η συνέχεια πολλές φορές είναι ελλειπής. Αυτό παντά νομίζω στην ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε. Η μελέτη αντικτύπου θα υποβληθεί στα μέλη του Κοινοβουλίου Επίσης όσον αφορά την Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ καλείται να κάνει μια συστηματική αξιολόγηση, έναν απολογισμό συστηματικό και τακτικό των δραστηριοτήτων της Όλαφ και αυτό βεβαίως το κάνει με μεγάλη επιμέλεια, προετοιμάζει γνωμοδοτήσεις για πολλά και διαφορετικά θέματα. Η Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ. Όσον αφορά την πλήρη αναρμόνιση των κυρώσεων, των ποινικών κυρώσεων, διασυνοριακά, οι ελάχιστες ποινές, Αυτά είναι σημαντικά θέματα και βεβαίως θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι αναφερόμαστε στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν εδώ προτείνει την υιοθέτηση μιας οδηγίας που θα επιβάλλει τις ελάχιστες ποινές και μία εναρμόνιση των κυρώσεων για την παραβίαση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τομείς του ποινικού δικαίου, πρόκειται για πράξεις αξιόπινες. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσης, τα πλαστά ευρώ, την επιβολή των ελάχιστων ποινών για αυτά τα αδικήματα και στην Ευρωζώνη, όπως ξέρετε, Σύμφωνα με την συνθήκη, το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η εναρμόνιση αυτών των ελάχιστων κυρώσεων και ποινών και η κοινή αντιμετώπιση ενός αδικήματος σε όλα τα κράτη-μέλη είναι κάτι που πρέπει να αφορά όλους μας. Ο κύριος Σοντή αναφέρθηκε στις αξιόπινες πράξεις που καλύπτει αυτή εδώ η πρόταση. Όχι μόνο απάτη, αλλά και άλλες παράνομες δραστηριότητες όπως νομιμοποίηση κονδυλίων που προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα, διαφθορά. Κάθε μορφή απάτης συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την οδηγία για την πλήρη προστασία των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ευρύ φάσμα λοιπόν ε, αξιόπινων πράξεων και όσον αφορά τη συνεισφορά, τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, πρέπει να σας πω ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ε, ήδη συμμετάσχει σε αυτήν την διαδικασία. Έχουν υποβάλει παρατηρήσεις έχουν εκφραστεί. Έχουν επεξεργαστεί την πρόταση και έχουν υποβάλει παρατηρήσεις. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προετοιμασίας έχουν εκφραστεί και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα επαναλάβω όμως για άλλη μια φορά ότι βεβαίως μπορούμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω το κείμενο και βεβαίως συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας και βεβαίως υπάρχει ένα κομμάτι εθνικής αρμοδιότητας Ο ΦΠΑ σαφώς αποτελεί τμήμα αυτής της οδηγίας στα έσοδα, στην πλευρά των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του προϋπολογισμού. Και για το θέμα της ανάγκης εναρμόνισης σε διασυνοριακό επίπεδο, σε σχέση με τους περιορισμούς. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από θεωρητικής απόψεως, αλλά στην πρόταση αυτή, στην οδηγία αυτή, προτείνουμε να εναρμονιστούν οι ελάχιστες Και όσον αφορά το καθεστώς των περιορισμών, η επιμήκυνση παραδείγματος χάρη των ε, ποινικών διαδικασιών με σκοπό να αποφευθεί η επιβολή ποινής ε, κύρωσης. Εδώ η επιβολή των ελάχιστων ε, περιορισμών για την πραγματική προστασία και αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που θα πρέπει να το επεξεργαστούμε περαιτέρω. Όσον αφορά τον Γενικό Εισαγγελέα. Εδώ βεβαίως υπάρχει μία βασική πρόταση όσον αφορά την ύπαρξη και τη δραστηριότητα αυτού του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα επεξεργαζόμαστε ακόμα περισσότερο την πρόταση αυτή και θα επανέλθουμε πολύ σύντομα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές με μια πιο εμπεριστατωμένη πρόταση. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο νομοθετικό κείμενο, μια φιλόδοξη πρόταση οδηγίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπεριέχει και την πρόταση για τον Ευρωπαίο ε, Εισαγγελέα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ε, τον Επίτροπο. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, βεβαίως θα συνεχίσουμε την συζήτηση της νομικής βάσεως ε, και διμερώς όσον αφορά το πολιτικό χρονοδιάγραμμα. θα πρέπει να το μάθουμε, να δούμε και πότε είναι ο καταλληλότερος χρόνος να περάσει το θέμα στην Ολομέλεια. Αλλά Είμαστε εδώ, ανταλλάσσουμε απόψεις ε, με τον αρμόδιο επίτροπο και ε, αξιολογούμε πολύ θετικά τις απαντήσεις ε, που λάβαμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Σεμέτα για την οδηγία ΠΥΦΕ. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τώρα την κοινή συνεδρίαση Κοντ Λίμπε και αμέσως να ξεκινήσουμε μάλλον να συνεχίσουμε με τη δική μας συνεδρίαση. so that will be the last. Shall I? Okay. Yeah, ladies and gentlemen. Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε με την συνεδρίασή μας από τις 9 ε, και 25 μέχρι τις 11.30 είχαμε μια πάρα πολύ έντονη ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή της Όλαφ. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα, αναπάντητα ερωτήματα όσον αφορά την παρέτηση του πρώην Επιτρόπου Ντάλι. Θελήσαμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Θα συνεχιστεί όμως το θέμα αυτό και σήμερα το απόγευμα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της Όλαφ για το 2012. Οι έρευνες ε, της Όλαφ και η διαμάχη μεταξύ αφενός του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ και της Επιτροπής Εποπτείας από την άλλη. Ο κύριος Τίμεμαντς, ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής Εποπτείας, αλλά και ένα άλλο ε, μέλος ε, της Επιτροπής Εποπτείας έχουν δηλώσει ότι αποχωρούν. Υπάρχουν λοιπόν δύο κενές θέσεις. Αυτή είναι η κατάσταση αν θέλετε. Κύριε Επίτροπε, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ και σας έχουμε ξαναζητήσει η Επιτροπή ως θεματοφύλακα των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει το ρόλο της. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την εξέταση του θέματος αυτού. Κύριε επίτροπε θα σας δώσω το λόγο για κάποια εισαγωγικά σχόλια και κατόπιν θα ζητήσω από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων αλλά και από τα μέλη της Επιτροπής να κάνουν τις παρατηρήσεις τους. Κύριε Σέμετα, έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Mr. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να ξεκινήσω με μια διευκρίνηση όσον αφορά την κατάσταση με την ε, Επιτροπή Εποπτείας. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί πλήρως η Επιτροπή Εποπτείας. Όλα τα μέλη ε, τα οποία έχουν ε, φύγει, έχουν αντικατασταθεί, λειτουργεί πλέον η Επιτροπή πλήρως και είναι σε θέση να λειτουργήσει ε, κανονικά και να καλύψει τα καθήκοντα τα οποία ε, οφείλει να καλύψει λόγω βάση της ε, νομοθεσίας. Υπάρχουν κάποια ζητήματα όσον αφορά την στρατηγική της Κομισιόν και τη θέση της Κομισιόν. Πριν αναφέρω συγκεκριμένα στοιχεία, θα ήθελα να σας πληροφορήσω για τις ε, εξελίξεις ε, μετά την ε, τελευταία μας συνάντηση της αρχής Μαΐου. Μετά τη συνάντηση 8 Μαΐου λοιπόν, πρότεινα στο Γενικό Γραμματέα της, Γενικό Διευθυντή συγγνώμη, της Όλαφ, ε, να ε, ε, υπάρξει μια κοινή συνεδρίαση με την Ερμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου με τη δική μου παρουσία έτσι ώστε να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση όσον αφορά την συνέχιση, το follow-up της Επιτροπής Εποπτείας σε σχέση και με την ετήσια έκθεση. και υπάρχει και ένα προσχέδιο οδικού χάρτη που περιλαμβάνει 17 συγκεκριμένες απτές δράσεις. Βάσει των συστάσεων της εκθέσεως της Επιτροπής Εποπτείας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πλέον οδεύουμε σταθερά και με επικοδομητικό τρόπο προς την υλοποίηση των συστάσεων ε, μέσα σε ένα πνεύμα συναντήληψης ε, όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει και το χρονοδιάγραμμα ε, υλοποίησης των συστάσεων. πρότεινα να γίνει η συζήτηση αυτή τη 12η Ιουνίου, αλλά δυστυχώς η Επιτροπή Εποπτείας δεν ήταν σε θέση να συμμετάσχει εκείνη την ημερομηνία σε μια τέτοια συνεδρίαση και θεώρησε πρόημο το γεγονός, δηλαδή θεώρησε πρόημη μια ενδεχόμενη συζήτηση. Εξακολουθώ πάντως να πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με τρόπο επικοδομητικό, γι' αυτό λοιπόν στόχος μου είναι, πρόθεσή μου είναι να διοργανωθεί μια τέτοια συνεδρίαση ε, τον Ιούλιο ή εν πάση περιπτώσει πριν από την διακοπή ε, για τις καλοκαιρινές διακοπές έτσι ώστε να υπάρχει αξιολόγηση των μέτρων και του οδικού χάρτη ε, και βεβαίως των μέτρων που θα πρέπει να υλοποιηθούν έτσι ώστε να υπάρχει όπως είπα και προηγουμένως συναντήληψη για τις δράσεις οι οποίες είναι και τις ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι συστάσεις της Επιτροπής Εποπτείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο τα μέλη της Επιτροπής, η κυρία Γκρέσλε από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Επίτροπε. Να σας πω καταρχήν ότι εδώ και ένα χρόνο ασχολούμαστε με το θέμα της Επιτροπής Εποπτείας και του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Αν κοιτάξει κανείς το κοινό σχέδιο δράσης, αυτό που μας στείλατε, Εγώ πραγματικά εδώ και εβδομάδες και μήνες ασχολούμαι με το θέμα αυτά και αυτό το κοινό σχέδιο δράσης εγώ θα συμφωνήσω εδώ με τον Γενικό Διευθυντή ότι υπάρχει μια προσπάθεια παρεμποδισμού του Γενικού Διευθυντή από μέρους της Επιτροπής Εποπτείας. Ε, θα αναγκαστώ να συμφωνήσω διαβάζοντας αυτό το κοινό σχέδιο δράσης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτή η Επιτροπή Εποπτείας δεν παρουσιάζεται σωστά και ότι αξίζει κάτι παραπάνω. Πρόκειται για ένα όργανο το οποίο έχει διοριστεί έτσι ώστε να υπάρξει μια παρακολούθηση, μια εποπτεία της Όλαφ. Δεν είναι εύκολη εργασία. Κύριε Επίτροπε, πάρτε το πολύ σοβαρά αυτό το θέμα και κάντε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει, να εργαστεί καλύτερα αυτή η Επιτροπή Εποπτείας. Πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και αν η Επιτροπή Εποπτείας ζητάει κάποια στοιχεία θα πρέπει να τους το δίνουμε. Είναι πολύ παράξενο το ότι μονίμως επικαλούνται την προστασία κάποιων δεδομένων. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι ήδη ο υπεύθυνος για την προστασία των στοιχείων από μέρους της Όλαφ είχε χρησιμοποιήσει αυτές τις δικαιολογίες, αυτές τις απαντήσεις για να παρεμποδιστεί η απόδοση συγκεκριμένων στοιχείων που είχαν ζητηθεί. Το ερώτημα λοιπόν όσον αφορά την ε, Επιτροπή Εποπτείας είναι πολύ σημαντικό και βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών που πρέπει εσείς να κάνετε. Πρέπει να σας πω επίσης ότι απορώ πάρα πολύ όταν είδα σε αυτήν την έκθεση τα όρια, τα κατώτατα όρια για τις απάτες. Παραδείγματος χάρη στο γεωργικό τομέα πρέπει να ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο ευρώ η απάτη για να ασχοληθεί η Όλαφ. Μα δεν είναι δυνατόν να βασιστούμε σε μια τέτοια στρατηγική καταπολέμηση της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν. Η πολιτική μου ομάδα δεν μπορεί να στηρίξει κάτι τέτοιο. Σήμερα το πρωί Ακούσαμε επίσης και κάποιες άλλες παρατηρήσεις όπως η αποστολή ή μη αποστολή κάποιων στοιχείων, κάποιων εγγράφων στις εθνικές αρχές ή υπερσυγκέντρωση κάποιων στοιχείων από την Όλαφ. Πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή Εποπτείας σίγουρα θα πρέπει να παίξει το ρόλο της. Ένα ρόλο διαβούλευσης. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το ότι η Επιτροπή Εποπτείας εγγυάται, βάζει ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε οι διαδικασίες να ε, γίνονται απρόσκοπτα. Αυτό νομίζω ότι εννοούμε εδώ. Και με ποιο τρόπο η Όλαφ υλοποιεί αυτές τις ε, διαδικασίες, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει εσάς σαν επίτροπο να σας απασχολήσει. Υπάρχουν 80 υποθέσεις παραδείγματος χάρη, οι οποίες δεν πέρασαν από την Επιτροπή Εποπτείας, οι οποίες εστάλησαν κατευθείαν στις εθνικές αρχές. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω πώς εσείς ε, αντιλαμβάνεστε τη βελτίωση αυτών των διαδικασιών και το ρόλο της Επιτροπής Εποπτείας. Και κάτι άλλο. Εμείς στείλαμε ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό το ερωτηματολόγιο έμεινε αναπάντητο στο 50% αυτών των ερωτήσεων. Πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε γιατί έμειναν αναπάντητες πολύ σημαντικές ερωτήσεις όπως 43, 45, 63, 67, 51, 50, β, α, 66, 75 μέχρι 77. Θα σας τα δώσω και γραπτά. Αλλά θεωρώ πραγματικά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί εδώ με την ε, διαδικασία αυτή που ξεκίνησε το Κοινοβούλιο γιατί δεν είναι δυνατόν να στέλνουμε ένα ερωτηματολόγιο, να στέλνουμε τόσο σημαντικές ερωτήσεις, οι οποίες παραμένουν αναπάντητες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος. Μια ολόκληρη δέσμη ερωτήσεων ακούσατε. Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Well, so I... Μάλιστα. Νομίζω ότι στην εισαγωγή μου αναφέρθηκα πολύ ξεκάθαρα σε αυτό και είπα ότι είναι προς το κοινό συμφέρον ε, του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Συμβουλίου η Όλαφ και η Επιτροπή Εποπτείας της να εργάζονται αποτελεσματικά. Γι' αυτό αυτό το σχέδιο δικού χάρτη υποβλήθηκε από εμένα και στην Επιτροπή Εποπτείας και στον Γενικό Διευθυντή της Όλαφ. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κυρία Γκρέσλε πως ε, για να συζητήσουμε κάτι κάποιος θα πρέπει να θέσει κάποια ε, θέμα, να θέσει το, τη βάση της συζήτησης επιτάπητος. Και αυτό το έγγραφο ήταν για έναν αρχικό προβληματισμό και σε επίπεδο Επιτροπής Εποπτείας, όλα και σε επίπεδο Γενικού Διευθυντή, όλα για την κατάσταση γενικώ και την εφαρμογή διαφόρων συστάσεων. Ελπίζω τον Ιούλιο να γίνει και μια συνάντηση όπου και οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους και να κατανοήσουν τα προβλήματα, που φυσικά και υπάρχουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, και κατάλαβα καλά αναφερθήκατε στην πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και management system. αλλάζει η κατάσταση. Όπως με ενημέρωσε ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής Αποπτίας, η Επιτροπή Αποπτίας αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται την αξιολόγηση των αναγκών της, των αναγκών της Επιτροπής Αποπτίας δηλαδή, ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσματική πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ε, ε, ρυθμίσει εργασία ένα έργο το οποίο υπέγραψε ο, πρώην πρόεδρος, ε, ο τέος πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας και προς της ε, Γενικός Όλαφ και από ό,τι με ενημέρωσε και η Όλαφ με την ισχύει αυτή η διευθέτηση, αυτή ο διακανονισμό, αλλά εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ή να ε, βελτιωθεί ο διαγωνισμός αυτός, θα υποβάλει τις προτάσεις φυσικά, τις ιδέες της. Ελπίζουμε το στομότερο δυνατόν και μετά ε, θα δούμε. Εμείς είμαστε, μάλλον η όλα φαντάζομαι ότι είναι ανοιχτή για αυτή σε κάθε πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της Επιτροπής Εποπτείας. Πάντοτε βέβαια με πλήρη σεβασμό στο, στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε στα κατόφλια, στα κατώτατα όρια. Μάλλον υπάρχει παρανόηση στην προηγούμενη συνάντησή μας προσπάθησα να, σε, να σας εξηγήσω τι εννοούμε. Εδώ δεν μιλάμε για κατόφλια. Με τους νέους κανόνες της Όλαφ θεσπίστηκε το σύστημα των λεγόμενων προτεραιοτήτων ε, στην πολιτική έρευνας. Investigative Policy Priorities. Αυτές οι προτεραιότητες βασίζονται σε τέσσερα κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνεται η αρχή της αναλογικότητας, όταν δηλαδή μπορούμε να έχουμε μια επιστροφή μετά η προστέμενη αξία που μπορεί να φέρει η έρευνα της Όλαφ σε σχέση παραδείγματος με το να αφαιθεί το έργο αυτό στις εθνικές αρχές, τρίτον η αποτελεσματική χρήση των πόρων της Όλαφ και τέταρτον υπάρχουν και ειδικά κριτήρια όπως είναι ο οικονομικός αντίκτυπος μιας υπόθεσης κτλ. Άρα υπάρχουν ποσά που αναφέρονται που δείχνουν τη σοβαρότητα της ε, υπόθεσης σε ένα δεδομένο τομέα. Αλλά αποτελούν ενδείξεις μόνο και για ένα μόνο από τα τέσσερα προαναφερθέντα κριτήρια. Σε ό,τι αφορά τώρα την πράξη, τις δραστηριότητες της όλα αυτές καθεαυτές, θα σας ξαναπώ ότι μετά το Φεβρουάριο του 12, οπότε και τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες, το 46% των υποθέσεων που ήταν ανοιχτές για τον τομέα των τελωνίων και των διαδοτικών ταμείων, αναφέρομαι, είναι ή, το κάτω του ορίου, του να ή έχουν άγνωστο οικονομικό αντίκτυπο. Το 46% λοιπόν Σχεδόν το ίμιση των υποθέσεων δηλαδή που είχαν ανοίξει ήταν κάτω από το 1 εκατομμύριο. Επίσης, όταν μιλάμε για προστασία των οικονομικών συμφέροντων της Ένωσης και για τη δραστηριότητα της Όλαφ, θα ήθελα να πω ότι το 2012 185 υποθέσεις άνοιξε Όλαφ στους δύο αυτούς τομείς σε σχέση με 82 το 2011, 59 το 2010 και 25 το 2009. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι, θεωρείτε ότι η αύξηση των υποθέσεων στον τομέα αυτό, μιλάμε για επταπλάσιες υποθέσεις σε σχέση με το 2009, είναι κάτι λάθος. δεν είναι μια ε, σωστή συμπεριφορά τη όλα. εγώ νομίζω ότι συνιστά μια σημαντική βελτίωση τη δραστηριότητα τη όλα, στου τομεί αυτού, του συγκεκριμένου. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενημέρωση της Επιτροπής Εποπτείας για τις αποθέσεις που έχουν κλείσει. Πρέπει να σας πω για μια ακόμη φορά ότι τουλάχιστον ε, με βάση τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, η Όλαφ τηρεί τους κανόνες που σχετίζονται με την υποβολή των πληροφοριών στην Επιτροπή Εποπτείας και αυτό πριν η υπόθεση σταλεί στις Εθνικές Δικαστικές Αρχές. Ο κανονισμός της Όλαφ δεν προβλέπει, δεν λέει ότι όλα πρέπει να περιμένει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εποπτείας για την υπόθεση που έχει κλείσει. Η Όλαφ τηρεί απαραίτητα τις απαιτήσεις του κανονισμού. Καταλαβαίνω ότι κατανοούμε διαφορετικά τον κανόνα αυτό. Από νομικής όμως πλευράς είναι νομίζω σαφές και στην υπόθεση η Φραντσέζικα αυτό καθάρισε και το δικαστήριο ότι δηλαδή όλα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας πριν στα υπόθεση στις Εθνικές Αρχές. Νομίζω ότι αντιλαμβάνει, γνωρίζετε τον κανονισμό. Έχουμε το άρθρο 11.1 του κανονισμού της Όλαφ που λέει πολύ ξεκάθαρα ότι ουδή συμπεριλαμβανομένη επιτροπή αποκτία ε, μπορεί να παρέμβει σε μια μονομένη έρευνα. Έτσι έχουν κανόνες. Έρχομαι στο ερώτημα για τα ποσοστά ποσοστά απαντήσεων. Θέλω να είμαι σαφής και σε αυτό το σημείο. Η Κομισιόν εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να σας δώσει τα πλήρη στοιχεία για να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις ε, διαδικασίες σε εξέλιξη. Δικαστικές μία στη Μάλτα, μία στο Λουξεμβούργο και μία στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά την υπόθεση Φρανσμπικ. οι Ο Φρανσέ ήταν ο τευτής της Eurostat, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, τότε τέλος πάντων, και η Κομισιόν έχασε αυτή την υπόθεση, κυρίως γιατί απεφάνθη το δικαστήριο ότι η αποκάλυψη Κομισιόν πολλές πληροφορίες. Και έτσι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθότητας. Κυρία για ένα λεπτό το πολύ να κάνει άλλη μια ερώτηση. Είναι γνωστό ότι σήμερα οι διάφορες υποθέσεις μπαίνουν σε κατηγορίες, σε πακέτα αν θέλετε είναι επίσης γνωστό ότι μετά από 18 μήνες κλείνουν τα διάφορες, οι διάφορες υποθέσεις στην Όλαφ. Και οι περισσότερες στατιστικές αυτές είναι διακοσμητικές. Τουλάχιστον εγώ αυτό ξέρω. Κύριε Επίτροπε. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω με αυτά που είπατε. Φεβρουαρίου του, συγγνώμη, 2012 τέθηκε σε ισχύ νέοι κανόνες και βάσει αυτών η Όλαφ ε, προχώρησε σε αξιολόγηση όλων των ε, υποθέσεων που έλαβαν χώρα σε διάφορες ε, και πρέπει να πω ότι πριν τη μεταρρύθμιση υπήρξαν υποθέσεις οι οποίες έμειναν ε, στο στάδιο της αξιολόγησης για πολλά χρόνια και αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Η Όλαφ λοιπόν προχώρησε, ε, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και ε, πήρε αποφάσεις για όλες αυτές τις υποθέσεις βάσει των νέων κανονισμών και ξανά και υποθέσεις για τις οποίες υπήρχε σοβαρή υπόνοια απάτης. Και επομένως αξιολόγηση έγινε για όλες τις υποθέσεις αυτές ε, τις λεγόμενες backlog. Ε, η Όλαφ λοιπόν θέλησε να αντιμετωπίσει όλες αυτές ε, τις υποθέσεις για τις οποίες, και, και οι υποθέσεις για τις οποίες ε, δεν απεδείχθη ε, με σαφήνεια το αδίκημα ή η παράβαση, αυτές ολοκληρώθηκαν, έκλεισαν. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θετικό και μάλιστα το θετικό του πράγματος αναγνώρισε και η Επιτροπή Εποπτείας. Εάν δεν σφάλω, σε πολλές περιπτώσεις ε, της ε, εκτίσης ΠΥΦ δεν ήταν ικανοποιημένο το Κοινοβούλιο με τις μακροσκελείς ε, διαδικασίες που σχετίζονται με το άνοιγμα παλαιών υποθέσεων. Και πρέπει να σας πω ότι Το 2011 ο μέσος όρος ε, ήταν 6,8 μήνες και τώρα είναι 1,4 μήνες. Και η γενική διάρκεια της ε, ερευνητικής ε, διαδικασίας από 29 μήνες το 11 έφτασε στους 6 μήνες το 12. Ε, στοιχεία τα οποία σαφώς καταδεικνύουν την βελτίωση των καταστάσεων και ε, το γεγονός ότι οι νέοι κανονισμοί βάσει των οποίων λειτουργεί η Όλαφ έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Και κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με την Όλαφ και τη διοίκησή της ε, υπογραμμίζω ακριβώς ε, αυτό ε, το θέμα ε, διορθώνω από 26 μήνες το 11 σε 22, από 29 μήνες 11 σε 22,6 μήνες το 12 και αναφέρω λοιπόν κάθε φορά σε επαφές μου με, το, με την Όλαφ ότι 22,6 μήνες είναι πολύ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που μας δίνει τη δυνατότητα με την παρουσία του να συνεχίσουμε να συζητάμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και τα προβλήματα με την όλα αυτή την Επιτροπή Εποπτείας και γενικότερα το όλο θέμα αυτό. Συγκεκριμένα θέλω να ρωτήσω, γιατί υπάρχουν αμφιβολίες. Ως Επίτροπος Αρμόδιος για την καταπολέμηση της απάτης, πότε μάθατε ότι ήταν υπό έρευνα ο κύριος Ντάλι ο συνάδελφός σας δηλαδή, για μια υπόθεση απάτη. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να μου πείτε πότε πληροφορηθήκατε το σχετικό. Επίσης, επειδή είναι ένα στοιχείο σύγκρουση συμφερόντων και ανησυχεί και μας ανησυχεί και εμάς κοινή γνώμη. Το 2004, από το 2004 μάλλον, ξέρετε ότι υπάρχει μια σημαντική συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων πολυεθνικών στον τομέα των καπνών και τη, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά ή μάλλον για να πω καλύτερα, για τη χρηματοδότηση ενός μεγάλου ε, τμήματος ε, των προγραμμάτων καταπολέμησης ε, του λαθρεμπορίου καπνού. Οπότε ξέρω, η Όλαφ ε, διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία αυτή. Ήταν κατά κάποιο τρόπο εκπρόσωπος μας με την νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις αυτές για τη συμφωνία. Πώς, με ποιο τρόπο λαμβάνει τελικά η Όλαφ χρηματοδότηση, τέλος πάντων συμμετέχει, ενέχεται στις συμφωνίες με τις ε, μεγάλες ε, τροπνοβιομηχανίες. Είδα μία δική σας ε, συνέντευξη, δεν ξέρω με ποια καπνοβιομηχανία τέλος πάντων. Ε, επειδή δεν μας τα καλά ο κύριος Κέσλερ πριν, θα ήθελα να δω αν μπορείτε εσείς να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Τρίτον, σε σχέση με την Επιτροπή Υποπτίας. Εσείς πώς αντιλαμβάνεστε την προστασία του οργάνου αυτού που για μας είναι πολύ σημαντικός και για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της όλα αφενός αλλά και κυρίως για τη διατήρηση της αξιοπιστίας της ως οργανισμού από τη φύση του προβληματικού που είναι απαραίτητος αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε ένα εισαγγελέα από την άλλη όμως. Προβληματικό ε, οργανισμό υπό ποια έννοια. Ε, στην αρχή εγώ είχα θέσει το ζήτημα του κώδικα διοντολογίας. Ότι η Όλαφ είναι ανάγκη από την αρχή να προασπίζεται τα συμφέροντα ε, του υποέρευνα ατόμου. Είτε είναι είτε δεν είναι ένοχος, ε, γιατί αν δεν είναι έχουμε την περίπτωση του κυρίου Νταλή, παρετείται, μετά αποδεικνύεται δεν είναι, πέντε μέρες μετά, τρία χρόνια μετά δεν έχει σημασία. Για την κυρία Σέμπρη τώρα, ε η οποία φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο είναι αντικείμενο σύγκρουση συμφερόντων, διότι ήταν η Μαλτέζα ε, εκπρόσωπος μέσα σε μια επιτροπή που όμως ε, ερευνούσε ζητήματα που αφορούσαν τη Μάλτα. Πώς ε, λύθηκε το πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων της κυρίας που ήταν σε κάποιες συνεντεύξεις, σε κάποιες ανακρίσεις, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος ήταν ο ρόλος της. Και σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε ούτε αυτό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να απαντήσετε αμέσως, αν συμφωνείτε. Uh, λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα, σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε ότι εγώ ως Επιτροπός είμαι υπεύθυνος για θέματα ε, πολιτικής, στρατηγικής και όχι για τις συγκεκριμένες ε, διαδικασίες ε, διαρεύνησης με τις οποίες δεν αναμειγνύομαι. Πληροφορήθηκα την για την παρέτηση του ε, Επιτρόπου Νταλή από τον πρόεδρο Μπαρόσο την ημέρα της παρετήσεώς του. Ήμουν μάλιστα στην Ινδία και ε, έλαβα σχετικό τηλεφώνημα από τον πρόεδρο που με πληροφορούσε για αυτό το συγκεκριμένο συμβάν. Tobacco issues uh, Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα του καπνού και, συμφωνία, και τη συμφωνία για τα προϊόντα καπνού. Πρέπει να κατανοήσουμε ποιος είναι ο ρόλος και το έβρος αυτής της συμφωνίας για τα προϊόντα καπνού. Ε, περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις για τις ε, μεγάλες καπιονοβιομηχανίες οι οποίες έχουν υποχρέωση ε, να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν όλα τα συστήματα ανείχνευσης track and trace των πακέτων τους. Υπάρχουν και κάποιες γενικότερες συμφωνίες όσον αφορά το tracking and tracing. και περιέχονται άρρωστε ε, και στην ε, οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμίσουμε. Είναι ένα μέτρο εξαιρετικά ε, σημαντικό που συμβάλλει στην καταπολέμηση και της παραχάραξης των προϊόντων καπνού αλλά και στην μείωση της λαθρεμπορίας των ιδίων η εφαρμογή των συστημάτων ε, ιχνηλασιμότητας, tracking and tracing, έχουν μειώσει κατά 30% το πρόβλημα στην, ε, στα πέντε χρόνια. Επίσης ε, υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες όσον αφορά τα κατασχεμένα τσιγάρα των αντίστοιχων μαρκών. Δηλαδή, Εφόσον κατασχεθούν ε, τα τσιγάρα αυτά πρέπει η βιομηχανία να πληρώσει και κάποια πρόστιμα ε, από την πλευρά των κρατών μελών. Επομένως, ε, τίθεται ένα σύστημα, ας πούμε, κώδικα συμπεριφοράς και τα χρήματα προσμετρώνται στο προπολογισμό των κρατών μελών και είναι σημαντικά ποσά. Γιατί και οι τέσσερις συμφωνίες, δηλαδή με τις τέσσερις ε, ε, εταιρείε <coughs> αντιπροσωπεύουν δύο δις το χρόνο στους προπολογισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρήματα αυτά δεν ε, πηγαίνουν απευθείας στην Όλαφ, πηγαίνουν στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν βλέπουμε να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την ε, συμμετοχή της Όλαφ στις διαπραγματεύσεις ε, με τις καπνοβιομηχανίες, γιατί ένας από τους ρόλους της Όλαφ είναι ακριβώς να βρίσκει τους τρόπους ε, και τα εργαλεία τα οποία θα δώσουν την ε, ε, μεγαλύτερη, τη μέγιστη ε, δυνατότητα καταπολέμησης της παραχάραξης των προϊόντων και επομένως πιστεύω ότι αυτές οι συμφωνίες ακριβώς δίνουν κάποια εργαλεία, ορισμένα από τα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Πρόσφατα είχαμε και νέα στρατηγική όσον αφορά το λαθρεμπόριο των ε, ε, τσιγάρων γιατί πιστεύουμε ότι ε, τούτο εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με την μέγιστη δυνατή σοβαρότητα και επομένως και η στρατηγική που αφορά το ζήτημα αυτό πρέπει να είναι εξίσου σοβαρή. Τώρα, όσον αφορά την Επιτροπή Εποπτείας, αναφέρατε και την λέξη προστασία. Νομίζω ότι στη συνάντηση της 28ης Μαΐου διαβεβαίωσα το σώμα ότι υπάρχει η ίδια μεταχείριση και προς την Όλαφ ε, και προς την Επιτροπή Εποπτείας. Και στην ίδια την Επιτροπή Εποπτείας τον Μάιο Ε, είπα ότι με μεγάλη σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε τις γνωμοδοτήσεις τους και τις συστάσεις τους ε, γιατί αποτελεί ένα πάρα πολύ, μια πάρα πολύ θετική ε, και απαραίτητη συμβολή input για την εργασία της Όλαφ. Επομένως, μεταξύ των δύο σωμάτων πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία. Ε, με, την, ε, σαφή, με το σαφή διαχωρισμό βεβαίως ότι και τα δύο σώματα είναι απολύτως ανεξάρτητα. Ε, πρότεινα λοιπόν τριμερή διάλογο και με δική μου δηλαδή συμμετοχή έτσι ώστε να διαλευκανθούν και κάποια ε, ζητήματα και να βρεθεί ο βέλτιστος δυνατός τρόπος υλοποίησης των συστάσεων της Επιτροπής, αυτές που παρουσιάζει στην ετήσια έκθεσή της η Επιτροπή Εποπτείας ε, γιατί ε, γίνονται οι προτάσεις και αν το σχέδιο δράσης συγκριθεί, πρέπει να υλοποιηθεί κιόλας. Και επομένως ε, η Όλαφ μαζί με την Επιτροπή Εποπτείας θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία ήλεγξαν. Ευχαριστώ πολύ και καθότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και έχουμε μόνο 10 λεπτά. Μια σύντομη συμπληρωματική ερώτηση είναι. Ευχαριστώ. Υπάρχει και στις δηλώσεις της Όλαφη Κομισιόν ότι η Όλαφ διαπραγματεύεται με τις καπνοβιομηχανίες στο πλαίσιο της συμφωνίας και θέλω να ξέρω Ποιο είναι το περιεχόμενο τη διαπραγματεύση αυτή, γιατί αν κατάλαβα καλά, διαπραγματεύεται εξ ονόματο τη Κομισιόν η Θέλετε να μα ε, διευκρινίσετε περί τίνο ακριβώ ε, πρόκειται, τι διαπραγματεύεται, το περιεχόμενο, τα προγράμματα, τι ακριβώ. Στα statements τη Κομισιόν και τη Όλαφ λέγεται, τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ, ότι διαπραγματεύεται ω εκπρόσωπο τη Κομισιόν η Όλαφ. Πρώτα, ευχαριστώ που τήρησα το χρόνο. Μια σύντομη απάντηση από τον Επίτροπο. Για να αποσαφηνίσουμε τη συμφωνία αυτή και τη λειτουργία της ε, συμφωνίας. Ήδη το 2004 ε, υλοποιήθηκε η πρώτη συμφωνία με την πρώτη δηλαδή ε, εταιρεία. Ο ρόλος της Όλαφ στη διαπραγμάτευση αυτών των συμφωνιών ήταν η παροχή πραγματογνωμοσύνης και γνώσεων. Γίνουν πιο αποτελεσματικές συμφωνίες αυτές. Έλαβα και επιστολή από τον κύριο Τόιερ έτσι ώστε να υπάρξει πρόσβαση στα έγγραφα της διαπραγμάτευσης. Ζητήσατε να ε, έχετε την δυνατότητα να συμβουλευτείτε, να μελετήσετε τα έγγραφα αυτά σε ένα ασφαλές ε, ε, δωμάτιο, σε, σε μια ασφαλή αίθουσα, έτσι ώστε τα μέλη της Επιτροπής, τα μέλη του Κοινοβουλίου ε, να μελετήσουν ε, στους χώρους του Κοινοβουλίου τα έγγραφα αυτά. Η άλλη τώρα. κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την υπομονή σας και για την παρουσία σας βεβαίως. παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια την Όλαφα, από όταν δηλαδή άρχισα να είμαι μέλος στην Επιτροπή Κόντουρ. Το πρόβλημά μου ήταν όχι αυτό που κάνει, αλλά αυτό που δεν κάνει η Όλαφ. Παρακολούθησα από κοντά και όλη αυτή την υπόθεση Νταλή. Και έχω την αίσθηση ότι υπάρχει, ε, ελοχεύει κατά κάποιο τρόπο μία ε, χαμηλής εντάσεως διαφωνία. Και μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι συνδυάστηκαν αυτά τα δύο στοιχεία, ε, οδηγώντας την Όλαφ σε πλήρες αδιέξοδο. Έχει εγκλωβιστεί η Όλαφ στην υπόθεση Νταλή. Έχουμε δεκάδες εκατομμύρια, ίσως οπωσδήποτε 20 εκατομμύρια δωροδοκίες στο, στο δημόσιο τομέα των χωρών. Ορισμένες χιλιάδες αφορούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια Ε, σε 40% των περιπτώσεων έχουμε ε, ανάκτηση. Εν πάση περιπτώσει έχει φτάσει σε αδιέξοδο η Όλαφ. Ερωτώ, τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε θεσμικά τουλάχιστον να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο αυτό. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς έτσι ώστε να μας οδηγήσετε πέρα από το αδιέξοδο αυτό. Πρόεδρος, ε, σύντομη ερώτηση, μήπως να έχουμε και μία σύντομη απάντηση. Το Επίτροπο Σέμετα. Πρώτα απ' όλα, η Όλαφ συνεχίζει τις ε, δραστηριότητές της. Και βλέποντας τα ποσά και τα αριθμητικά στοιχεία, βλέπετε, θα διαπιστώσετε, ότι στη διάρκεια του 12 υπήρξε εντατικοποίηση των προσπαθειών. Το 2012 λοιπόν η Όλαφ είχε πάνω από 1.700 ε, ε, περιπτώσεις επιλεγμένες ε, έναντι 900 περίπου τον προηγούμενο χρόνο και ακόμα λιγότερον το 10. Επομένως βλέπουμε ότι έχει υπερδιπλασιαστεί το ποσοστό. Και αυτό δείχνει ότι η Όλαφ ε, αισθάνεται άνετα με αυτήν τη μεταρρύθμιση και τους νέους ε, κανόνες και δουλεύει αποτελεσματικότερα από ό,τι στο παρελθόν. Όσον αφορά την ε, πολιτική δράση, τη στρατηγική δράση που χρειάζεται, πρέπει να πω ότι πρώτα πρέπει να εγκριθεί, να εγκριθούν μάλλον οι τροποποιήσεις του κανονισμού Όλαφ, να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των αρχών γιατί ε, με τον τρόπο αυτό διευθετείται το ρυθμιστικό πλαίσιο από διάφορες σκοπιές και αυτή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό ζητήσαμε το Κοινοβούλιο να ε, ασχοληθεί και να ψηφίσει για το θέμα αυτό, για την οδηγία αυτή, στην επόμενη Ολομέλεια του Στρασβούργου. Εφτά χρόνια κράτησαν οι διαπραγματεύσεις ε, για την πρόταση αυτή. Κρίμα θα ήταν να μην είμαστε σε θέση να επιτύχουμε συμφωνία όσον αφορά αυτό το τελικό στάδιο. Κατά τα λοιπά, είναι σημαντικά και αυτά που είπα και στην προηγούμενη, απαντώντας στην προηγούμενη ερώτηση δουλεύουμε εντατικά για τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για ποινικού χαρακτήρα διερευνήσεις. Θα, ε, αντιμετωπιστούν ξέχωρα πλέον αυτές οι περιπτώσεις από τις ε, διοικητικές διαδικασίες και θα υπάρχει πλέον ένα ισχυρό εργαλείο ε, για να αντιμετωπιστούν οι ποινικώς προλάσιμες πράξεις οι οποίες αφορούν το οικονομικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την έγκριση της ε, οδηγίας μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τον ε, κανονισμό και να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο κάποιες από τις πρόνοιες. Σκεφτόμαστε ας πούμε και το ενδεχόμενο να εισάγουμε ένα σύστημα ανεξάρτητου ελεγκτή για τις, ε, ε, που θα ε, εγγυάται για, την σωστή, για τις σωστές διαδικασίες και που θα βλέπει το θέμα και από τη σκοπιά των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη δράση στρατηγικής και βεβαίως από αυτού θα πρέπει να υπάρξει ιδέουσα διαβούλευση και με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο έτσι ώστε το νομοθετικό πλαίσιο ε, για την Όλαφ να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό. Uh, uh, Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Δεν είναι καν ερώτηση, είναι μια συμπληρωματική παρατήρηση. Το θέμα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα είναι πολύ σημαντικό εδώ, γιατί πολλές φορές ε, αναγκαζόμαστε να κάνουμε τέτοιου είδους ε, προτάσεις. Το συντομότερο δυνατόν λοιπόν παρακαλώ πολύ κάνετε αυτή την πρόταση. Η πράσινη. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κανείς δεν σας ζητά να παρέμβει η Επιτροπή Εποπτείας στις διερευνήσεις της Όλαφ. Όμως, εσείς πρέπει να εγγυηθείτε την αξιοπιστία της Όλαφ, η οποία πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι επικρίσεις που ακούγονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον πρόεδρο, από την σημαντικότερη πολιτική ομάδα, που ζήτησε την παρέτησή του. Και το ίδιο και η ομάδα μου. Σήμερα το πρωί μας είπε ο Γενικός Διευθυντής ότι μπορούμε να το ζητήσουμε όσες φορές θέλουμε, εκείνος δεν πρόκειται να παρατηθεί γιατί προστατεύει την ανεξαρτησία της Όλαφ. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι σήμερα το πρωί στην ακρόαση και πιστεύω ότι γνωρίζετε τι συνέβη, διαπιστώσαμε ότι ένας υψηλόβαθμος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ, ψεύδεται. Ψεύδεται τουλάχιστον σε ένα από τα ερωτήματα που μας απάντησε. Η κυρία Σόνμπρι, επικεφαλής της ομάδας για την καταπολέμηση της απάτης της Μάλτας, συμμετείχε σε μία συνάντηση και η απάντηση στην ερώτηση είναι όχι. Όταν του έκανα λοιπόν αυτή την ερώτηση σήμερα, είπε ναι τουλάχιστον σε τρεις συνεντεύξεις. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ψέμα λοιπόν αυτό που μας έστειλε γραπτά. Τουλάχιστον ένα ψέμα. Αν λοιπόν κύριε Σέμετα καλούσαμε εδώ έναν επίτροπο και διαπιστώναμε ότι ο επίτροπος ψεύδεται, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται ο Επίτροπος αυτός να είχε διοριστεί. Ο κύριος Κέσλερ ψεύδεται, είναι αποδεδειγμένο αυτό που σας λέω. Δεν είναι υπόνοια ούτε υπόθεση. Προτίθεστε να ξεκινήσετε μία πειθαρχική διαδικασία κατά του κυρίου Κέσλερ. Ναι ή όχι. Εμείς δεν τον καταδικάζουμε. Ζητάμε πειθαρχική διαδικασία και να μπορέσει να μας απαντήσει. Πρόκειται για κάποιον ο οποίος ήρθε εδώ και μας είπε ψέματα. Ε, ε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση. Ε, Uh, <laughs> uh, uh, λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί με ακρόαση και εμείς πρέπει να αναλύσουμε τα αποτελέσματα αυτής της ε, συζήτησης. Οι υπηρεσίες μου ενημέρωσαν ότι Δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσει. Και άμα λάβετε υπόψη α, β, γ, δ και τα λοιπά υπό ερωτήσεις, ήταν πάνω από 200 οι ερωτήσει. Πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν έπρεπε να συνταχθούν οι απαντήσει. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα αυτό που έθεσε στο Κοινοβούλιο, και σας λέω τι με ενημέρωσαν, τι μου είπαν. Το θέμα ήταν αν η κυρία Σκέμπρη είχε λάβει μέρος στην έρευνα. Η απάντηση ήταν ότι δεν συμμετείχε στην έρευνα, αλλά συμμετείχε ως διερμηνέας σε μια κρόαση επειδή ο μάρτυρας χρειαζόταν μετάφραση. Αυτή είναι η μέρωση που έχω. Θα δω βέβαια και θα μελετήσω το θέμα μόλις φύγω από εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμπληρωματική ερώτηση, ένα λεπτό. Κοιτάξτε, μπορούμε να παίξουμε αυτό το παιχνιδάκι εδώ και πολύ καιρό έχουμε ξεκινήσει. Ουσιαστικά δείχνεται αλληλεγγύη στην Επιτροπή. Ο Πίτερ Πολ Ζάμιτ αποφάσισε να εγκαταλείψει την υπόθεση του πρώην Επιτρόπου Ακούμε ότι πρόκειται για μία έρευνα η οποία δεν έχει καμία αξιοπιστία. Αν την είχα ε, ξεκινήσει εγώ θα με είχαν διώξει. Και ο κύριος Κέσλερ παίζει με τις λέξεις. Αυτό κάνει. Δεν είναι πρόκειτο για μία παρουσία για να μεταφράσει, για να κάνει τη διερμηνέα. Πρόκειται για συνέντευξη. Και η ερώτησή μου είναι σαφής, την επαναλαμβάνω. Κάποιος ο οποίος είπε ψέματα εδώ στο Κοινοβούλιο προτίθεστε να τον υποβάλλετε σε πειθαρχική διαδικασία. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. <laughs> Uh, uh, uh, Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι απλά να επαναλάβω τι μου είπαν πριν μπω στην αίθουσα αυτή. Ότι πρόκειτο περί παρερμηνίας, ε, παρανόησης της ερώτησης. Ε, ήταν ένα λάθος. Ελπίζω να το δέχεστε, να το καταλαβαίνετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά... τις δηλώσεις ενός εξωματικούς αστυνομίας, όχι ενός ε, στη Μάλτα. Ε, πρέπει να κάνουμε μια πολύ σαφή διάκριση μεταξύ της διοικητικής διαδικασίας, της διοικητικής έρευνας και της ποινική έρευνας. Η Όλαφ έχει αναλάβει τη διοικητική έρευνα. Η ποινική έρευνα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι σε εξέλιξη στη Μάλτα και αν διάβασα καλά την απομαγνητοφώνηση αυτού του αξιωματικού αστυνομίας ε, είπε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις. Και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω, στην προκειμένη περίπτωση. Πρόεδρος. Τελευταία πολιτική ομάδα, η ECR, όχι, με συγχωρείτε, διορθώνω η Γκου. Ο κύριος Ντεγιόν. Η Σερ δεν είναι παρόντες. Ντεγιόν. Δεν είμαι από την Γκου, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ενωτική Τέλος πάντων. Είχα κάνει μια ερώτηση νωρίτερα σε σχέση με την ποιότητα των ερευνών της Όλαφ, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτά που γίνονται στη Μάλτα και αυτά που ακούσαμε από τα κράτη-μέλη. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. αν ε, συμφωνήσουμε αυτά που λέει ο Επίτροπος, ε, ίσως αυτή η μελέτη που μας δώσει λίγο παραπάνω φως σε αυτή την κατάσταση. Ό,τι αφορά τώρα την Επιτροπή Εποπτείας, η οποία είπε ότι αν θέλουμε να ερευνήσουμε τι γίνεται σε μια μεμονωμένη υπόθεση ή δεν μας δίνουν έγγραφα ή αν μας δώσουν είναι έγγραφα που τα πιο πολλά τα έχουν σβήσει. Και πράγματι, ένα πολύ μεγάλο μέρος έκθεση έχει διαγραφεί, είναι ζησμένο. Το ίδιο βέβαια παθαίνουμε και εμείς όταν ε, κάνουμε ερωτήσεις, δεν παίρνουμε απαντήσεις. Και το μόνο επιχείρημα Γι' αυτό είναι, α, είναι θέμα προστασίας δεδομένων. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν αυτά τα στοιχεία που δεν παίρνουμε εμείς και η Επιτροπή Εποπτείας. Υπάρχει μια ομάδα σοφών, υπάρχει ε, μια επιτροπή να αναλάβει αυτό το θέμα, γιατί η πρόταση που κάνετε για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ενδεχομένως και για έναν εισαγγελέα Ευρωπαίο. Τι θα, αποτέλεσμα θα έχει για τη δουλειά της Όλαφ. Επίσης μας είπε ο Γενικός Διευθυντής ότι έχει αιτήματα από την Γενική Γραμματική, από τις, από τις Γενικές Διευθύνσεις να βάλει πιο ψηλά ε, στον κατάλληλο των προτεραιοτήτων κάποια θέματα και να τα δει πιο ε, γρήγορα. Συμφωνείτε για να όχι πρέπει να διακοπεί αυτή η πρακτική. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Κύριε Επίτροπε. Λοιπόν, θα απαντήσω στην πρώτη. Και να δώσω κάποια πιο πρόσφατα στοιχεία. 71 αιτήσει αυτή τη Συμβουλευτική Επιτροπή μετά την υιοθέτηση των νέων κανόνων και όλες αυτές οι αιτήσει για τις οποίες δόθηκε πλήρης πρόσβαση στις υποθέσεις. Στις 61 υποθέσεις από τις 71 και για τις υπόλοιπες δεν ζητήθηκε το δεύτερο στάδιο της πρόσφασης. Τώρα, όσον αφορά το γεγονός ότι έρχονται τα έγγραφα με κάποια ε, τμήματά τους ε, δυσανάγνωστα ή σβησμένα ή ελλειπή, Υπάρχουν συγκεκριμένες εντολές όσον αφορά αυτήν την πρακτική. Και οι συνεργάτες της Όλαφ γνωρίζουν τους κανόνες. Εγώ από πολιτικής απόψεως θα σας πω ότι εάν υπάρχουν επιπλέον δυσκολίες και προβλήματα στο σημείο αυτό, τότε θα πρέπει να επεξεργαστούμε εκ νέου τους ε, κανόνες λειτουργίας, να τους βελτιώσουμε. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε μια αμοιβαία κατανόηση μεταξύ της Επιτροπής Εποπτείας και της Όλαφ. Μην ξεχνάτε ότι εδώ αναφερόμαστε σε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες, λεπτές πληροφορίες και θα πρέπει οι κανόνες να είναι σαφέστατοι, κατανοητοί από όλους και όλα αυτά τα πολύ ευαίσθητα αν θέλετε στοιχεία και όλες αυτές τις πληροφορίες δεν μπορεί να δίνονται έτσι χωρίς καμία διαπίστευση και προστασία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο. Ε, βεβαίως ο ρόλος μου είναι να διευκολύνω αυτήν την ε, βελτίωση των κανόνων, να υπάρξει πλήρης σαφήνεια. Πλήρης σαφήνεια για το τι ισχύει μεταξύ Όλαφ και Επιτροπής Εποπτείας. Εγώ θέλω και οι δύο ανεξάρτητες αυτές αρχές, φορείς, να συνεργαστούν με τον καλύτερο τρόπο. Προτεραιότητες τώρα. Φυσικό είναι ο καθένας από εμά να θεωρεί ότι η υπόθεσή του, η περίπτωσή του πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν προτεραιότητα. Ο καθένας θεωρεί ότι η δική του υπόθεση είναι η πιο σημαντική. Αυτό που πρέπει εδώ να δούμε είναι ο διευθυντής της Όλαφ να παίρνει ανεξάρτητα αποφάσεις, να κάνει τη δική του εκτίμηση, εάν ναι ή όχι μια συγκεκριμένη υπόθεση είναι προτεραιότητα ή όχι. Και αυτός είναι και ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ την διεξαγωγή αυτών των ερευνών. Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσαμε όλους τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Γκρέσλε όμως έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Μπαλτσίτης. Πριν τους δώσω το λόγο, θα ήθελα σαν επικεφαλής αυτής της Επιτροπής να σας πω, κύριε Σέμετα, εκτιμάμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ήρθατε σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε και θεωρούμε πραγματικά ότι το θέμα αυτής της μεσολάβησης που έχετε αναλάβει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εποπτείας και της ΟΛΑΦ είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι σημαντικός ο ρόλος σας και είναι και σημαντική λειτουργία και συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο ανεξάρτητων φορέων. Τώρα, έρχομαι στο πιο δύσκολο τμήμα. Όταν σας αποστέλουμε ερωτήσεις σε εσά στην Επιτροπή και διαπιστώνουμε ότι οι μισές από αυτές είναι αναπάντητες, αυτό είναι τελείως ε, μη ικανοποιητικό, για να το πω έτσι. Έχουν ε, απαντηθεί πολλές ερωτήσεις, αλλά πολύ σημαντικές ερωτήσεις που έθεσε το Κοινοβούλιο παρέμειναν αναπάντητες, αγνοήθηκαν. Αυτό για μας είναι πραγματικά κάτι το πολύ απαξιωτικό και δείχνει ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας, να δημιουργηθεί ένα κλίμα δυσπιστίας μεταξύ μας. Σας ζητώ λοιπόν να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Πρόκειται για μια καθαρά διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τρίτον, όσον αφορά τις έρευνες Όλαβ για κάποιες περιπτώσεις διαφθοράς. Τον Οκτώβριο λοιπόν δόθηκε απαλλαγή και στην υπόθεση αυτής της στην οποία, η οποία μας απασχολεί σήμερα, συγγνώμη, οδήγησε τη, στην παρέτηση του Επιτρόπου από τη Μάλτα. Βλέπουμε ότι τουλάχιστον προσωρινά η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει γιατί διαπιστώθηκε ότι ο κύριος Ντάλι δεν είναι εμπλεγμένος σε αυτή την υπόσθεση διαφθοράς. Δεν αποδεικνύεται τουλάχιστον τίποτα τέτοιο από την μέχρι τώρα έρευνα. Πότε θα συζητηθεί λοιπόν και η πολιτική διάσταση αυτής της υπόθεσης. Θα περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου που έχει ξεκινήσει ο Επίτροπος Ντάλι. Γιατί τελικά είδαμε ότι η παρέτηση του κυρίου Ντάλι πλέον δεν έχει λόγο ύπαρξης. Μήπως θα πρέπει η Επιτροπή να αναλάβει το θέμα καθότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν και να υποστηρίζουν πλέον αυτήν την απόφαση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές άμεσα εκλεγμένοι από τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν σαν κύρια αποστολή τους ε, να προχωρήσουν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και αφού σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, αρκετή τεκμηρίωση για την υπόθεση του Επιτρόπου Ντάλι και μπορώ να σας υπενθυμίσω ότι πριν από εννέα μήνες η υπόθεση παρουσιάστηκε τελείως διαφορετική. Ακούσαμε τότε για πολύ σοβαρές ενδείξεις. Ε, βλέπουμε λοιπόν εδώ να υπάρχει πολύ μεγάλη αντίφαση από το πώς παρουσιάστηκε τότε η υπόθεση αυτή και τι αποδεικνύεται τελικά σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαντηθούν οι ερωτήσεις που σας στείλαμε. Δεν είναι μόνο υποθε... Ε, ερωτήσεις που αφορούν την υπόθεση Ντάλι, αλλά και άλλες υποθέσεις καταπολέμησης ε, της απάτης και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ενδεχομένως το πλαίσιο ε, το θέτει η υπόθεση Ντάλι. Η συνδιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι δεν θα κληθεί ο Πρόεδρος Βαρόζο. Εμείς σαν Επιτροπή Ελέγχου του Προεπολογισμού αναλάβαμε μετά από εντολή της συνδιάσκεψης των Προέδρων να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και να υποβάλουμε τα συμπεράσματά μας στην συνδιάσκεψη των Προέδρων, στις πολιτικές ομάδες και τέλος και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι εύκολη αυτή η αποστολή και το θέμα είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας αντιμετωπίζει σαν άξιος να διεκπαιρέσουμε αυτό το έργο και προτίθεται να μας υποστηρίξει, να μας βοηθήσει. So, uh, I think that, uh... Αυτό που πραγματικά μπορώ να πω είναι ότι αυτό που μόλις είπατε ισχύει η Κομισιόν προσπαθεί να έχει τη μέγιστη δυνατή διαλειτουργικότητα με το Κοινοβούλιο. Και εμείς απαντήσαμε στα ερωτήματα τα οποία έθεσε το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι όλοι κατανοούμε ότι η Ευρωπαϊκή ένωση είναι ένωση κράτους δικαίου. Και είναι πολύ σημαντικό το κράτος δικαίου να γίνεται δεόντως σεβαστό. Όταν η Κομισιόν απαντάει στις ερωτήσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντελεχώς αξιολογεί τις ε, απαντήσεις σε σχέση με την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Όταν υπάρχει ε, δικαστική διαδικασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε τρεις-τέσσερις τέτοιες ε, υποθέσεις και στο Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο. Τότε η Κομισιόν δυστυχώς δεν είναι σε θέση να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που τις έχουν τεθεί, διότι αφορούν αυτές τις ε, υποθέσεις, ε, οι οποίες δεν έχουν ακόμα τελεσιδικήσει ενώπιον των δικαστηρίων. Ε, θέλω να ζητήσω από το Κοινοβούλιο να κατανοήσει τη θέση αυτή. Κοιτάξτε και τις αποφάσεις του δικαστηρίου κατά το παρελθόν. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις ε, έχασε η Κομισιόν, αλλά στις περιπτώσεις τις οποίες έχασε, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν έγινε σεβαστό το τεκμήριο αθωότητος. Γι' αυτό ακριβώς η Κομισιόν προστατεύει και τον εαυτό της Έχουμε λοιπόν διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη ενώπιον των δικαστηρίων και επομένως ζητώ να κατανοήσετε ότι δεν μπορούμε να ενεργήσουμε διαφορετικά εμείς στην Κομισιόν. Είμαστε οι θεματοφύλακε των συνθήκων, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο, Διαδικαστικό, κύριο Στά, Κύριε Επίτροπε, ε, κοιτάξτε, δύο οι δύο αυτές νομικές υποθέσεις τις οποίες αναφερθήκατε τι σχέση έχουν με την Όλαφ. Έχουμε μία υπόθεση ενώπιον των βελγικών ε, δικαστηρίων. Έχουμε την υπόθεση Ντάλι κατά Swedish Match. Δεν έχει να κάνει με την Όλαφ αυτό. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι η Swedish ε, ε, Match ήρθε στην Επιτροπή και είπε διάφορα για τον Επίτροπο Νταλή. Δεύτερον, ε, δεύτερον, αμφισβητείται ο τρόπος με τον οποίο έλαβε χώρα η παρέτηση του Επιτρόπου Νταλή. Ε, δεν έχει να κάνει ούτε αυτή η υπόθεση με τις ε, έρευνες ε, της Όλαφ αφορά την ημέρα της 16ης Οκτωβρίου που εσείς από ό,τι μας είπατε είσαστε στην Ινδία. Τι σχέση... Αυτό είναι διαδικαστικό, γιατί ο, ο κύριος Επίτροπος απαντάει και οι ερωτήσεις του δεν είναι σωστές, οι απαντήσεις του συγγνώμη δεν είναι ορθές. Πρόεδρος, ε, ε, αναφερθήκατε σε δύο ε, υποθέσεις, όχι, είναι τρεις υποθέσεις. Η τρίτη είναι στην Μάλτα. Η νομική υπηρεσία της ε, Κομισιόν αξιολόγησε ενδελεχώς την κατάσταση. Και όσον αφορά τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των απαντήσεων για υποθέσεις οι οποίες ακόμα, των οποίων μάλλον οι δικαστικές διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή είναι η θέση της Κομισιόν. κυρία Γκρέσλη, ο κύριος Βαλδίτης και παρακαλώ να δοθεί μια κοινή απάντηση. Κύριε Πίτροπε, δεν μπορούμε εμείς να συμπεριφερόμαστε εδώ σαν ε, υπεύθυνοι ένοχοι για το ότι μπορεί ενδεχομένως να χάσει στο δικαστήριο την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Η παρέτηση Η ουσιαστικά οδήγησε σε μια συνέντευξη τύπου και ακολούθησαν 15 ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι οι συναντήσεις και κλεισμένων των θυρών. Εμείς κάνουμε τέτοιες συναντήσεις και κλεισμένων των θυρών, όμως είδαμε ότι οι δηλώσει στον τύπο και οι συνεντεύξεις ήταν η μία μετά την άλλη. Και αυτό που φυσικά ακολούθησε δεν έχει άμεση σχέση με αυτό που έκανε η Επιτροπή, γιατί η υπόθεση στο Λουξεμβούργο στο δικαστήριο έγινε μετά από πρωτοβουλία και προσφυγή του Επιτρόπου Ντάλι. Σας ερωτώ λοιπόν, πώς δικαιολογείται η έρευνα, η ελλειπής έρευνα της Όλαφ, γιατί σε αυτό βασίζεται τελικά η έλλειψη στοιχείων στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Και ρωτώ το να πηγαίνει κανείς και να γευματίζει με έναν πολύ σημαντικό μάρτυρας αποτελεί τμήμα της διαδικασίας της αποδεκτής και ο μάρτυρας ή ε, μάρτυρας είπε ότι είχε πιει, ότι την πίεσαν να πιει, τη βοήθησαν να μεθύσει. Αυτά τα είπε στο δικαστήριο. Δεν είναι φήμες. Επίσης κύριε Επίτροπε, όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν να κοιτάξει κανείς τους αριθμούς για το 2012 για την Όλαφ, διαπιστώνει ότι υπάρχουν τόσες πολλές περιπτώσεις οι οποίες δεν ολοκληρώνονται που βλέπουμε ότι πάνω από 400 υποθέσεις, 423 ε, υποθέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν και οι μισές από αυτές έκλεισαν μέσα στη διάρκεια του έτους. Μα δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για μείωση του χρόνου επεξεργασίας. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Είμαστε ίσως περιορισμένης νοημοσύνης ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά όχι τόσο περιορισμένης ώστε να μην μπορούμε να καταλάβουμε αυτούς τους αριθμούς. Εννοείται ότι έχουν παρουσιαστεί λανθασμένα στοιχεία. Και αυτό μπορεί να είναι μια υπόθεση απάτης. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Θα ήθελα να σας ε, ε, ζητήσω να μην με αγνοήσετε στο μέλλον, γιατί περίμενα πάρα πολλή ώρα μέχρι να μου δώσετε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο που ήρθε στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας και ελπίζω να μην ε, του κακοφανεί η σημερινή διαδικασία. Αυτό που συμβαίνει σήμερα ε, ε, βρίσκεται, συγκαταλέγεται στις υποχρεώσεις του Επιτρόπου η Όλαφ, η υπηρεσία της, η Επιτροπή Εποπτείας, ε, είναι όλα στοιχεία ε, και υπηρεσίες οι οποίες ε, βοηθούν την Κομισιόν αλλά και το Κοινοβούλιο βεβαίως να υπεραμεινθούν των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να καταπολεμήσουν την απάτη. Η Όλαφ και η Επιτροπή Εποπτείας μη λησμονούμε ότι χρηματοδοτούνται από τους ενωσιακούς πόρους. Επομένως, είναι υπόλογοι με την έννοια ότι πρέπει να λογοδοτούν οι οργανισμοί αυτοί για την διαχείρισή τους στις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Εποπτείας δεν ε, συμφώνησε να συμμετάσχει στην, ε, στην κοινή συνεδρίαση. Και εμείς αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε τι γίνεται εδώ. Καταλαβαίνουν το ρόλο τους εκεί στην Επιτροπή Εποπτείας, ναι ή όχι. Είναι δυνατόν να αρνείται η εποπτεία εποπτείας η Επιτροπή Εποπτείας ε, να αρνείται να ε, συναντήσει τον πολιτικό της προϊστάμενο. Η ανεξαρτησία της Όλαφ και η ανεξαρτησία της Επιτροπής Εποπτείας βεβαίως πρέπει να διασφαλίζονται. Πλην όμως αυτό παρασάγκας απέχει από το θέμα που μας απασχολεί εδώ ε, και από την διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων. Κύριε Επίτροπε, όταν υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ των διαφόρων οργάνων, πρέπει να βλέπουμε τι προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός. Και νομίζω ότι οι πρόνοιες είναι σαφείς και αναφέρονται στις τακτικές συνεδριάσεις οι οποίες δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Βεβαίως στη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων δεν θα γίνει λόγος για τις τρέχουσες διερευνήσεις προφανώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαλτσίτης. Λοιπόν, λέει ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν θα σταθώ στις ε, κατηγορίες ε, οι οποίες, ε, τις οποίες μου απευθύνατε, αλλά ξέρετε εδώ δίνουμε το λόγο στις πολιτικές ομάδες σύμφωνα με το μέγεθος. Το μέγεθος κύριε Μπαλσίτης πρέπει να σας πω ότι μετράει σε μερικές περιπτώσεις λέει ο Πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει όμως πέρα από τον αστεϊσμό ε, θα ήθελα να σας ζητήσω να με συγχωρέσετε. Δεν, ήταν καμία, δεν είχα καμία πρόθεση να σας αγνοήσω. Η κυρία Γιάλα Σέντερ από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Σύντομη να είστε παρακαλώ. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είμαι πολύ σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαμέτα για την παρουσία του εδώ, αλλά και να υπενθυμίσω ότι ως Επίτροπος είστε ένα είδος διαμεσολαβητή ε, μεταξύ δύο οργάνων που έχετε υπό την ευθύνη σας. Το ότι όλα και η Επιτροπή Εποπτείας λειτουργούν σωστά ε, είναι δική σας τον να λειτουργούν σωστά είναι δική σα ευθύνη κατά κάποιο τρόπο. Είναι πολύ πολύ πολύπλοκοι και σημαντικοί οργανισμοί. Πρέπει να του προστατεύσουμε. Εσεί είστε υπεύθυνο. Κάτι παραπάνω από μεσολαβητή. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί η υπόθεση αυτή ξεκίνησε όταν αποφάσισε όπως μας είπε ο κύριος Κέσλερ, να ξεκινήσει αφού άκουσε κάποιες ε, ε κυρίες, γκρέι κτλ. Ε, ξεκίνησε μια αντιπαράθεση με καλή πρόθεση ξεκίνησαν όλα ίσως, αλλά τώρα παίζεται το κύριο της Όλαφ. Εσείς είπατε ότι ενημερωθήκατε όταν παρετήθηκε ο κύριος Ντάλ Πάντως ε, ευθύνη έχετε, δεν είστε ένας απλός διαμεσολαβητής ε, και γι' αυτό ε, πρέπει να έρθετε να μας μιλήσετε στην Επιτροπή μας. Είναι σημαντικό και ο ρόλος σας αυτός πρέπει να διατηρηθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανεξαρτησία τη Όλαφ, ο κύριος Οντί Έκανε ε, μια ερώτηση στο Γενικό Διευθυντή της Όλαφ σήμερα το πρωί και του είπε ότι αν μεγαλώσει, αυξηθεί η έλλειψη εμπιστοσύνης ε, και τα ερωτηματικά σε σχέση με το χειρισμό της υπόθεσης και η Κομισιόν είπε ότι η Όλαφ είναι, γιατί η Όλαφ έδωσε στην Κομισιόν στοιχεία, έτσι ξεκίνησε. Μάλιστα μπορεί να λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Τέλος πάντων η Κομισιόν μας λέει λίγο πολύ αυτό. Αν λοιπόν αυξηθεί η δυσπιστία του κοινοβουλίου απέναντι στο πρόσωπο του κ. Κέσλερ, τον ρωτήσαμε, τον κύριο, κύριο Σοντή συγκεκριμένα, τι θα κάνει. Και είπε ότι πάνω απ' όλα, ε, ακόμη και από το Δημοκρατικό από το Κοινοβουλίο, τελικά βρίσκεται η ανεξαρτησία τη Όλαφ Και δεν θα παραιτηθεί. Εσεί συμφωνείτε, γιατί εμένα πραγματικά με σόκαρη απάντηση που έδωσε ο κ. Κέσλερ στην ερώτηση του κ. Σοντή Γιατί εγώ θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο είναι ε, αυτό που έχει τον τελευταίο λόγο τον έλεγχο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στην προκειμένη περίπτωση που δεν έχει σεβαστό τεκνοσαρθότητα, είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Συμφωνείτε με την άποψη του κ. Κέσλερ ότι είναι ακόμη πάνω και από το δημοκρατικό έλεγχο η ανεξαρτησία τη Όλαφ. Mm. Απάντησε ο επίτροπο για να καταλήξετε κύριε Επίτροπε, σας δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αν συμφωνείτε να απαντήσω στα ερωτήματα των αξιότιμων βουλευτών. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία, θέλω να διευκρινίσω ότι εγώ δεν είμαι στατιστικολόγος, είναι, είμαι οικονομολόγος στο επάγγελμα και όλα τα στατιστικά στοιχεία τα οποία μιλάμε έχουν δημοσιευτεί στην ετήσια έκθεση της Όλαφ για το 2012. Και θα μπορούσαν όλοι οι βουλευτές να αναλύσουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Δεν υπάρχει κανένας κρυμμένος κρυφός υπολογισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των απαντήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τις επιπτώσεις τα αποτελέσματα της έρευνας ή των δικαστικών υποθέσεων. Νομίζω πρέπει να είναι σαφές. Για να μην φτάσουμε σε τη δικασία κύρωσης ε, μεταξύ άλλων λόγω παράτυπων ερευνών της Όλαφ. Είναι ένα θέμα που μπορεί να σχετίζεται και με το αν απαντήθηκαν ε, εν το χρόνο κάποια ερωτήματα κτλ. κτλ. Είναι σημαντικό το θέμα, εμείς ε, το επεξεργαζόμαστε και βλέπουμε και τις απαντήσεις και μελετάμε και τις ε, εξέλιξη δικαστικές ε, ε, δικασίες. Θέλω να επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό το κράτος δικαίου να γίνεται σεβαστό. Αυτό ισχύει για την προκειμένη περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τη δρόση του κ. Μπαλτσίτης, θέλω να τον ευχαριστήσω για τις υποδείξεις του. Και πρέπει να σας πω, κύριε Μπαλτσίτη, ότι έχουμε τακτές ανταλλαγές απόψεων με την Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ και τον Γενικό Διευθυντή της Όλαφ. Και πράγματι προσπαθήσαμε να διοργανώσουμε μια κοινή συνεδρίαση μεταξύ Επιτροπής Εποπτείας, Όλαφ, και κομισιόν και ίσως καλό θα ήταν αυτό να γίνει μια τακτική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Όλαφ και Επιτροπής Εποπτείας και με τη δική μου συμμετοχή. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν εγκριθεί μεταρρύθμιση της Όλαφ θα παράσχει επιπρόσθετα μέσα και εργαλεία για την ε, βελτίωση του έργου της Επιτροπής Αποπτείας. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μία από τις διατάξεις αφορά την ανταλλαγή απόψεων σε πολιτικό επίπεδο. Σε σχέση με τις προτεραιότητες των δραστηριοτήτων της Όλαφ. Αυτό προβλέπεται στον κανονισμό της Όλαφ. Γι' αυτό και θεωρώ τόσο σημαντικό το ότι τελικά θα ήταν να καταλήγουμε σε συμφωνία για το σημαντικό αυτό θέμα. Τώρα για τη διαμεσολάβηση και τα λοιπά. Νομίζω ότι έχουν σχέση αυτά τα δύο ερωτήματα μεταξύ τους. Να πω πρώτα απ' όλα ότι θα ήταν σφάλμα η σχέση μεταξύ Όλαφ και Επιτροπής Εποπτείας να συσχετιστεί με την υπόθεση Νταλή. Διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι Όλαφ διενέργησε μια πολύ σημαντική εσωτερική μεταρρύθμιση σε αρχές του 2012 Όλες οι διαδικασίες αναθεωρήθηκαν, επανεξετάστηκαν, η οργανωτική δομή άλλαξε. με επικέντρωση πλέον στις έρευνες, είναι κάτι το οποίο είχε ζητήσει πολλές φορές το Κοινοβούλιο, αλλά και το ελεκτικό συνέδριο, με τις εκθέσεις του. Και βέβαια με την Επιτροπή Εποπτείας υπάρχει και αυτή να εργάζεται από τις 2012 φαίνεται ότι η μέθοδος εργασίας και η κατανόηση του ρόλου της Επιτροπής Εποπτείας είναι λίγο διαφορετικός. Μιλάω για την συγκεκριμένη, την ε, τωρινή επιτροπή της σχέση με την προηγούμενη. Και φυσικά χρειάζεται κάποιος χρόνος και από τις δύο πλευρές μέχρι ότου κατανοήσουν η μία την άλλη. Εγώ βλέπω ότι αυτή η διαδικασία ε, συνεχίζεται και βεβαίως ε, θα κάνω την μπορεί να τη διευκολύνω. Για να έχουμε δύο ανεξάρτητους φορείς που θα λειτουργούν αποτελεσματικά. Thank uh. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι έγινε σαφές πόσο σημαντικό και πόσο σοβαρό είναι για εμάς ευρωβουλευτές αυτό το θέμα. Χρειάζεται πραγματικά να έχουμε την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όχι μόνο θα απαντά στα πολύ έτσι, ειλικρινή ερωτήματα, ανοιχτά ερωτήματα, αλλά θα αναπτύξει και τη μελλοντική δομή για να έχουμε μία ε, αποτελεσματική στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και περιμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη ανταλλαγή απόψε. Members, we continue immediately with the next points. Συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο ευθύ αμέσω. So, uh, Ειδική έκθεση 17 και 18 σημεία της ημερήσιας διάταξης πρόκειται για τις ε, ειδικέ ε, ειδικές εκθέσεις και ζητώ από τον David Bostock από το Ελεκτικό Συνέδριο να μας κάνει επίσης την παρουσίασή του. Προηγουμένως όμως θα σας ε, ανακοινώσω τον τίτλο της πρώτης έκθεσης «Αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης» να δώσουμε αμέσως το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο. Ο κύριος Μπόστοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μπορώ να σας κάνω μια παρουσίαση της έκθεσης. Δεν χρειάζεται όμως αφού το έχετε το έγγραφο. Το έγγραφο του εισηγητή κάνει μια εξαιρετική σύνοψη αυτών που στείλαμε στην έκθεσή μας. Θα αναφερθώ σε δύο σημεία μόνο. Πρώτον, σελίδα 5, εδώ το έγγραφο αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής για ομάδες υποστήριξης της ποιότητας που κατάφεραν να ξεπεράσουν προβλήματα βιωσιμότητας που είχαμε εντοπίσει στην έκθεσή μας. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από μέρους της Επιτροπής, αλλά βεβαίως δεν είναι και πάρα πολύ πιστική. Δεν είναι πολύ πιστική γιατί, διότι πρώτα αυτές οι ομάδες υποστήριξης ποιότητας δεν αφορούν όλες τις δαπάνες και ότι παραδείγματο χάρη όσον αφορά τα θέματα παροχής πόσιμου ύδατος υπάρχουν βασικές ε, ελλείψεις. Ο έλεγχος όσον αφορά την βιωσιμότητα των προγραμμάτων, παράγραφος 44 της έκθεσης, δείχνει ότι δεν ήταν θεωρητικό το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν στην πράξη. Πώς λειτουργούν αυτές οι ομάδες υποστήριξης της ποιότητας, παραδείγματος χάρη. Και εδώ δεν έχουμε απάντηση και ο εισηγητής καλά έκανε και έχει προσθέσει το σημείο 8 στις συστάσεις του. Και τώρα σελίδα 6. Εδώ ξεπερνάμε το φάσμα του ελεγκτικού συνειδρίου, τις συστάσεις μας και τα πορίσματά μας. Το σημείο 5 αναφέρουμε ότι το θέμα δεν είναι ποια είναι η παροχή υπόσημου ύδατος για τα νοικοκυριά ή η παροχή ύδατος για την γεωργία. Η ουσία εδώ είναι ότι υπάρχει θέμα χρηματοδότησης και κάποιος θα πρέπει να πληρώσει. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Πρόεδρος, ο εισηγητής ή η Επιτροπή. Ο εισηγητής θέλει να ακούσει την Επιτροπή. Ωραία. Ποιος θα μιλήσει από την Επιτροπή. Πολ Ρινιέ λέγομαι. Ευχαριστώ πολύ. Προσεκτικά ανέλησε η Κομισιόν τα σχόλια και τις συστάσεις του εισηγητού ε, συνειδητοποιεί η Κομισιόν τα σημεία και καθώς επίσης και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω ε, ζητήματα για τις περιπτώσεις που αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Θα παράσχουμε πληροφορίες ε, ανά project για την παρούσα κατάσταση και για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί ή που πρέπει ακόμα να ληφθούν. Αναπερίπτωση. Εσωτερικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε για ένα χρόνο να παρακολουθεί ε, ε, τις ε, παρούσες διαδικασίες και να διασφαλίσει ότι λειτουργούν σωστά εμείς δηλαδή, εμείς εσωτερικά με τα εργαλεία που έχουμε στην ε, διάθεσή μας, συγκεκριμένα ε, για τα projects που αφορούν πόσιμο είδωρ, να κάνουμε αυτόν τον εσωτερικό έλεγχο. Εάν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει για μία ακόμα φορά ε, τις ιδιαίτερες καταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με την απάντησή μας στην έκθεση της του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που φαίνεται ότι δεν έχει λάβει επαρκώ υπόψη όλα τα στοιχεία του εγγράφου εργασία. Ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκη η πραγματικότητα επιτόπου. Επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο παραδείγματα τα οποία βρίσκονται εις το, στην έκθεση. Ένα μικρό πρόγραμμα στην Ιγυρία, μικρό πρόγραμμα παροχής ε, ύδατος. Θα πρέπει να ανατρέξουμε ε, 14 χρόνια πριν περίπου, γιατί αυτό ξεκίνησε το 2001 η Νιγερία μόλις ε, ε, βγήκε από μια κατάσταση ιδιαίτερης αναταραχής ε, και επομένως ξεκίνησαν προγράμματα γρήγορης υλοποίησης για την βοήθεια προς την Ιγυρία. Γνωρίζουμε πως έχουν ε, όλες αυτές οι χώρες που ε, ε, βρίσκονται σε περίοδο αμέσως μετά το τέλος μιας μεγάλης κρίσης. Βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο στην ουσία. Όταν πρέπει κανείς να ξεκινήσει ένα project, αλλά δεν υπήρχε, δεν διαχείριση, δεν υπήρχε διοίκηση, πρέπει να αρχίσει από το μηδέν. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Παρόλα αυτά, το 2003 ε, ξεκίνησε, προχώρησε το έργο. Ε, και ξέρετε πώς έχει η κατάσταση. Είναι η υπογραφή συν τρία χρόνια για να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος. Η εκτέλεση είναι δύσκολη επιτόπου. Είναι πολλαπλά τα προβλήματα και νομίζω ότι πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη. Αυτό που κάνουμε στην Ιγυρία επιπλέον είναι ότι από το 2004 δόθηκαν πάνω από 17 εκατομμύρια ε, για το νερό γενικότερα. Δηλαδή ένα συνολικότερο ποσό και 10 χρόνια αργότερα για να σας δώσω λίγο και τη γενική εικόνα για το πόσο δύσκολο είναι και πόσο μακρύ ε, ε, είναι, πόσο χρόνο παίρνει για να βελτιώσουμε αυτά τα συστήματα. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφέρω είναι η υπόθεση της Γκάνα, στη βόρεια περιφέρεια της Γκάνας. Πρέπει να σας πω ότι η περιφέρεια αυτή είναι μία περιοχή ε, εκεί που είχαμε ε, ε, μία μεγάλη αιστεία μόλυνσης. Επομένως προβληματική η περιφέρεια και επιπροσθέτως πρόκειται για μία περιοχή με ιδιαίτερα υδρογεολογικά προβλήματα. Επομένως τα προβλήματα είναι πολλά ε, και όταν κανείς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα άλλα υφιστάμενα υγειονομικά προβλήματα, ε, δεν πρέπει να εκπλήσεται κάποιος όταν ε, με αυτές τις προϋποθέσεις ότι δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί. Το ξέραμε αυτό από την αρχή, αλλά μπορούμε να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει αιστεία μόλυνσης ε, σε αυτήν την ε, περιφέρεια της Γκάνας. Και αυτό είναι πολύ καλό. Ε, επομένως τα πράγματα δεν είναι η άσπρα ή μαύρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να εστιάζουμε την προσοχή μας στα γενικότερα αποτελέσματα γιατί ξέρετε δεν αρκεί κανείς να πει τόσα νοικοκυριά θα έπρεπε να έχουν πόσιμο νερό, ε, τόσα έχουν τελικά, άρα αυτό είναι προβληματικό. Πρέπει να ε, ε, έχει κανείς μια γενικότερη εικόνα σε λίγο βάθος χρόνου. Εγώ δουλεύω πάρα πολλά χρόνια σε αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες και έρχομαι συχνά συνέχεια σε επαφή με τους παρόχους ε, νερού και με τους εμπλεκόμενους και αυτό είναι πιο εύκολο να το λέει κανείς παρά να το κάνει. Ε, υπάρχει ένα διτό σύστημα. Έχουμε και την αποκέντρωση, αποκεντρωμένη διαχείριση, διακυβέρνηση, περιφερειακές κυβερνήσεις, κεντρικές κυβερνήσεις. Όλα αυτά για να δρομολογηθούν ε, παίρνει χρόνο. Δεν θέλω να βρίσκω δικαιολογίες, απλώς λίγο να ξαναβάλουμε τα πράγματα στη σωστή στόχευση. Μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία αποφασίστηκαν από το 2001 μέχρι το 2007. Τώρα είμαστε στο 2013 και βεβαίως η Κομισιόν έμαθε πολλά από τα λάθη και από το παρελθόν. Επομένως, ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι και εμείς ε, ε, πλέον ε, έχουμε πιο βελτιωμένη προσέγγιση όσον αφορά την επικεντρωμένη διαχείριση, όσον αφορά τα τιμολόγια. Έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα συζήτησης, συνδιαχείρισης, αλλά αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος. Επίσης προχωρήσαμε και εσωτερικά γιατί γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν οι απαραίτητοι έλεγχοι ποιότητας ε, και αξιολογήσεις κινδύνου και ε, συστήματα ε, εποπτείας. Εδώ έγινε αναφορά σε μια συγκεκριμένη ομάδα χριστών. Quality Support Group System. Αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο έχει δώσει αποτελέσματα, έχει βελτιώσει ε, διάφορα ε, έργα. Έχουμε δύο τέτοιους ελέγχους, ε, ένα, δύο ελέγχους στη διάρκεια των προγραμμάτων. Έχουμε επίσης ε, και την εποπτεία η οποία σχετίζεται με την χρήση των ε, πόρων. Ξεκίνησε δειλά, έχει τώρα ανδρωθεί, αλλά δεν είναι αρκετά δυνατό σύστημα. Επίσης, αυτή τη στιγμή συζητάμε με τη Γενική Διεύθυνση ΑΦΚΟ για τις δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης ε, αυτού του συστήματος Ρώμα, όπως το ονομάζουμε. Ε, έτσι ώστε να μην έχουμε μονάχα ένα monitoring ε, σε κάποια στιγμή του προγράμματος, αλλά ε, συγκεκριμένο monitoring, συγκεκριμένη οπτία για το κατά πόσον οι συστάσεις έχουν ακολουθηθεί. Um, and... Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία ήθελα έτσι να υπογραμμίσω ε, οπωσδήποτε τις συστάσεις τη διαβάσαμε προσεκτικά ε, οπωσδήποτε θα έχουμε την απαραίτητη διάδραση και για τα 23 έργα Τώρα μας ζητάτε και αναφορά, ενδεχομένως εδώ αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες. Αυτό που θέλουμε ε, να καταθέσουμε είναι ότι κατανοούμε ότι από υγειονομικής απόψεως και όσον αφορά, τις αποχετε... Ε, και όσον αφορά ε, τις υποδομές αποχέτευσης πρέπει να υπάρξει περαιτέρω προσπάθεια έτσι ώστε ε, και το τμήμα των υποδομών αποχέτευσης να είναι πιο αντιπροσωπευτικό. Ευχαριστώ. Ο συγητής Μπαρτστάς, κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Ναι. Όχι. Ο συγήτής. Νομίζω ότι αφού ακούσαμε αυτό που μας είπε το Ελληνικό Συνέδριο, και τα έγγραφα, δεν έχουν από πολλά. Ας ακούσουμε καλύτερα την Κομισιόν, θα ήταν χρήσιμο πιστεύω. Να δούμε αν τελικά υπάρχει προθυμία να γίνουν αυτά που ζητάμε στην παράγραφο 8 και 9. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλες μέθοδοι. Για το θέμα τη υδροδότηση ή της αποχέτευσης μπορούμε να εξετάσουμε τη διατύπωση για να είναι λίγο πιο έντονη και για να συμπεριλάβουμε τα σχετικά στην πολιτική μας. Όποιος έχει πάει επί τόπου, βλέπει και καταλαβαίνει τα πράγματα. Στην πρώτη μου παράγραφο μιλάω ειδικά για το πρόγραμμα της Βόρειας Νιγηρίας, Closing the Gap Ίσως όμως θα μπορούσαμε να είμαστε πιο σε, ε, ξεκάθαροι στη διατύπωσή μας για όσους χρειαστεί να διαβάσουν αυτό το κείμενο αργότερα και για τον εισηγητή που θα είναι πάνω για την διαδικασία απαλλαγή. Να κάνουμε δηλαδή επικοδομητικές ε, παρατηρήσεις. Yeah, ε. vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι Αν ο κύριος Μπόστοκ θέλει να ξαναπάρει το λόγο, η Επιτροπή μπορούν, όχι. Ωραία. Επόμενη έκθεση. Κύριε Μπόστοκ, πρόεδρε, και εδώ τι να σας πω. Το έγγραφο του κύριου Στάς είναι μία σαφέστατη σύνοψη της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Συμφωνεί η Επιτροπή με τις συστάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτή τη φορά θα περιοριστώ σε δύο σημεία των συστάσεων, το σημείο 7 των συστάσεων που ξεπερνάν την έκθεση και τις προτάσεις της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Το σημείο 4 πρέπει να σας πω εδώ ξαφνιαστήκαμε στο ελεγκτικό συνέδριο όσον αφορά την συντήρηση των δρόμων που πρέπει να γίνει από τοπικές επιχειρήσεις. Ναι, η συντήρηση σε καθημερινό επίπεδο, αν θέλετε, όντως γίνεται από τοπικές επιχειρήσεις. Όμως, μία περιοδική τακτική συντήρηση, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό στην παράγραφο 19 της έκθεσης, αναφέρομαστε σε αυτήν την συντήρηση που γίνεται από τοπικές επιχειρήσεις ενώ υπάρχει πρόβλημα εμπειρίας, τεχνολογίας, αποτελεσματικότητας αυτών των επιχειρήσεων. Ξαφνιαστήκαμε λοιπόν από αυτό το σημείο 4 πώς προτείνεται εδώ. Ευχαριστώ ο η Επιτροπή. Θέλετε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να επαναλάβω ότι η έκθεση Αγγλικού Συνεδρίου είναι πρόσδεκτη. Κατά μια θετική έκθεση αν δεν δούμε και το περιεχόμενο, το, συγγνώμη, το πλαίσιο, Αφρική, άρα πολλέ αντισώμενες χώρες, καταλαβαίνετε ότι τα βορίσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Και στι έξι χώρες ε, που έγιναν επισκέψεις ότι ε, παρατηρούνται βελτιώσει και αυτό είναι θετικό. Οι περισσότεροι οι περισσότεροι δρόμοι ε, ε, ήταν σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι πολύ καλό, σε ποσοστό πάνω από 90% τώρα. Ξεκολουθούν να διακυβεύονται πολύ σημαντικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε την ε, τακτική συντήρηση και την περιοδική, τη συντήρηση ρουτίνας και την περιοδική συντήρηση. Ξέρουμε ότι όταν ε, κατασκευάζεται ένας δρόμος, κατασκευάζεται για μια περίοδο 50 ετών. Αυτό σημαίνει ότι την 7η-8η χρονιά ξανακατασκευάζεται το οδόστρωμα. Και τα επόμενα χρόνια γίνεται μόνο συντήρηση. Καθαρίζεται δηλαδή το δικό δίκτυο και όλα αυτά τα... Ναι, τέλος Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι περιοδική στήριξη και συντήρηση ρουτίνας είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα διαφορετική μεθοδολογία, διαφορετικέ δεξιότητε απαιτούνται. Η Κομισιόν λοιπόν τι έκανε, τι κάνει σε όλα αυτά τα προγράμματα. Προσπαθεί όσο το δυνατόν περισσότερο να συμμετάσχουν οι τοπικέ μικρομεσαίες επιχειρήσει που αυτέ καλούνται να φέρουν σε πέρα τα έργα συντήρηση ε, του δικού δικτύου στην περιοδική συντήρηση, όταν χρειάζεται βαρύς εξοπλισμός, είναι πιο, δύσκολες, πιο δύσκολα τα έργα. Εκεί χρειάζεται σίγουρα μεταφορά τεχνογνωσίας. Σε πολλές περιπτώσεις στην Αφρική, ξένες εταιρείε αναλαμβάνουν το έργο αυτό, σε πολλές περιπτώσεις. Θέλω επίσης να αναφέρω κάτι που δεν φαίνεται ξεκάθαρα στην έκθεση του ελληνικού Συνεδρίου. Όταν μιλάμε για Paved Network και road, Roads Visited. Αν λάβουμε υπόψη μας μόνο δρόμους που έγιναν πριν από, λιγότερο από πριν από 8 χρόνια, το ποσοστό αυτό που είναι κάτω των πολύ, καλών, πολύ καλής κατάστασης ε, ε, σε άποψη αντιστοιχούν στο 58%. Σε αυτούς τους δρόμους η συντήρηση ρουτίνας γίνεται αποτελεσματικά. Εμείς δεν μιλάμε για τα προβλήματα στο μείζον δίκτυο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Κομισιόν, αλλά για, μιλάμε για ερωτικούς δρόμους μικρότερους δρόμους που βλέπουμε σε αφρικανικές χώρες. Η απάντηση που δώσαμε λοιπόν στη σύσταση του εισηγητή είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών έργων και μπορούμε μεταξύ μέσα σε αυτά τα έργα να προωθήσουμε τις ε, τοπικές εταιρείες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε σιγά σιγά να αναλάβουν την εκτέλεση αυτών των έργων. Ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και τι απαραίτητε ε, υποδομέ capacity building. Σύσταση παριθμών 7. Εκπώνηση έκθεση ή υποβολή έκθεσης με το τι κάνει η Επιτροπή σε θέματα πολιτικής και συγκεκριμένα για το περιβάλλον ε, και την ε, προώθηση της οδικής ασφάλειας. Υπάρχουν πολλά μέτρα που εφαρμόζουμε, όπως είπαν ε, οι συνάδελφοι για τα έργα έδρευσης, υδροδότησης. Έχουμε ένα πρόγραμμα στο επίπεδο για την ποιότητα, στο επίπεδο της μελέτης και του σχεδιασμού του σχεδίου θέλουμε να υπάρχει και ένα είδος περιβαλλοντικού screening σε κάθε project. Όπου χρειάζεται πλήρης περιβαλλοντική επίπτωση ή αλλιώς μπορεί να χρειάζεται να μελετηθούν κάποια περιβαλλοντικά μέτρα. Διαχωρίσουμε τα σχέδια δηλαδή σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Σε επίπεδο της αντιπροσωπείας γίνεται αυτό screening. Στο επίπεδο τώρα της υλοποίησης του project, φροντίζουμε να υπάρχει πάντοτε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το πεντάστη στη σύμβαση και είτε ο ίδιος εργολάβος, είτε κάποια μη κυβερνητική οργάνωση, κάποια τοπική αρχή το αναλαμβάνει. Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν τα περιλαμβάνουμε σε αυτή την εργαλειοθήκη που έχουμε για το προσωπικό μας που εργάζεται στα προσωπία, τα εξηγούμε όλα. Αν η συγκητή θεωρεί ότι είναι χρήσιμο θα μπορούσαμε να εκπονήσουμε ένα μικρό σημείο με όλα αυτά τα μέτρα, να δώσουμε και κάποια παραδείγματα, τι εντολές δίνουμε δηλαδή στο προσωπικό, τι οδηγίε δίνουμε στο προσωπικό τη αντιπροσωπία και στον ομόλογο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής, ο κύριος στα Ik wist natuurlijk dat, uh, dat de punten 4 en 7... Πρόεδρε, ήξερα ότι το σημείο 4 και το σημείο 7 θα προκαλέσουν ε, αντιδράσεις. Κατά κάποιο τρόπο ξεπερνούν, αν θέλετε, και το γνωρίζω αυτό, την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι όμως και ο ρόλος μας να προσθέσουμε μια πολιτική διάσταση. Σημειώνω αυτά που ανέφερε η Επιτροπή όσον αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου των υποδομών και εγώ πήγα στην Αφρική και είναι πάρα πολύ οδυνηρό να διαπιστώσει κανείς ότι ξένοι εργαζόμενοι, ξένες εταιρείες αναλαμβάνουν τα έργα. Λες και δεν υπάρχει αρκετή γνώση, εμπειρία και εργασία επιτόπου. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο. Για μεγάλα έργα υποδομής, οι ξένες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν πολλές φορές τα έργα. Και εγώ ήμουν παρόν σε μια τέτοια περίπτωση έργων υποδομής στο Κονγκό με κινέζικες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή αντέδρασε με πολύ ενδιαφέρον τρόπο και άκουσα πολύ προσεκτικά αυτό που είπατε, να μας δώσετε δηλαδή και τα στοιχεία και τις οδηγίες που δίνετε επί τόπου. Μπορείτε να μου στείλετε ένα μικρό σημείωμα. Δεν θέλω όλο το κείμενο για να μπορέσω να είμαι πιο συγκεκριμένος και εγώ. Ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεσή της. Ήταν εξαιρετική και αυτή και η προηγούμενη. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος άλλος Θέλω να πάρει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, δεν βλέπω κανένα. Κύριε Μπόστοκ από το ελεγκτικό συνέδριο, τι έχετε να προσθέσετε τίποτα. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 13, το οποίο το είχαμε αναβάλει. Δυστυχώς ο εισηγητής ε, δεν μπορεί να είναι παρόν, έχει ένα οικογενειακό πρόβλημα. Μπορούμε όμως να δώσουμε το λόγο στο ελεκτικό συνέδριο και θα λάβει υπό, ε, η συζήτηση χώρα μια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Μελέτησε το ελεγκτικό συνέδριο τις άμεσες ενισχύσεις για τους ε, ε, κτηνοτρόφους ε, θυλαζουσών αγελάδων, προβατίνων και εγών. Γνωρίζετε ότι ο κύριος στόχος αυτών των ενισχύσεων είναι να διατηρηθεί η παραγωγή σε περιοχές που δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ε, και επομένως ε, ε, γίνεται, διατηρείται αυτή η ενίσχυση ανα, ε, αναζώο έτσι ώστε να διατηρηθεί η οικονομική δυνατότητα της περιοχής. Ε, όλα τα, ε, ε, οτιδήποτε ξεφεύγει από το decoupling της βοήθειας είναι κατεξαίρεση. Έγιναν λοιπόν κάποιες εξαιρέσεις και τα κράτη-μέλη είχαν την δυνατότητα ε, να ζητήσουν εξαίρεση από την αρχή του decoupling και επομένως ε, να ε, ζητήσουν εξαίρεση που ονομάστηκε εξαίρεση μερική για το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων. Και αυτό έγινε για τις Τιλάδες, τις Αγελάδες, τις Προβατίνες και τις Αίγες. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι νομοθετικού περιεχομένου προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ΚΑΠ για την περίοδο 2012-2020 δίνει την δυνατότητα να συνεχιστούν αυτές οι ρητές βοήθειες σε ορισμένους παραγωγούς και στη νέα ε, χρηματοδοτική περίοδο. Παρόμοιες λοιπόν ενισχύσεις θα ε, είναι δυνατόν να συνεχιστούν μετά και το 2013. Τρία σημεία θα με απασχολήσουν όσον αφορά τις παρατηρήσεις του συνεδρίου. διεπίστωσε το ελεγκτικό συνέδριο ότι οι ενισχύσεις αφορούν το σύνολο της ενωσιακής επικρατείας και ουχή μόνο τις περιοχές ε, στις οποίες εξ αρχής θα έπρεπε να περιοριστούν και όπου επομένως αυτή η εντατική κτηνοτροφία είναι θεμελιώδου σημασίας για την οικονομική επιβίωση της περιοχής. Ε, επομένως, συστήνει το ελεγκτικό συνέδριο καλύτερη στόχευση της ενίσχυσης ε, και ζητά από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω των ε, επιδοτήσεων, συγγνώμη, των ενισχύσεων αυτών ε, που θα συνεχιστούν και για την περίοδο 2014-2020. Οι τρόποι καταβολής της ενίσχυσης ε, προφανώς θα αναφερθούν στις κατεξα... La cour πράξης. Επίσης λέμε ότι οι ενισχύσεις αυτές ε, αποτρέπουν σοβαρές οικονομικές ε, αρνητικές ε, επιπτώσεις, οικονομικές, κοινωνικές και κτηνοτροφικής παραγωγής. Εμείς όμως διαπιστώσαμε ότι η, την, αυτή η μορφή κτηνοτροφίας δεν είχε σχέση ούτε με το coupling ούτε με το decoupling και απλώς σε κάποιες ιδιαίτερες περιοχές όπως ας πούμε η Σκοτία και η Πορτογαλία τελικά οδήγησε σε μείωση του ζωικού ε, κεφαλαίου και σε μείωση της εκτεοτροφικής παραγωγής. Συστήνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή, το ελεγκτικό συνέδριο το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη να καθορίσουν τις πιο σημαντικές δραστηριότητες ε, καθώς επίσης και τις περιφέρειες οι οποίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Επ' αυτού η Κομισιόν ε, απεφάνθη και απήντησε ότι αυτό αποτελεί κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Συμφωνούμε, πλην όμως θεωρούμε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καθορίσει τους τρόπους με τους οποίους ε, δεσμεύονται τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τις ενισχύσεις αυτές στα πλαίσια των ε, ε, μέτρων που έχουν ληφθεί ήδη στην αναθεωρημένη ΚΑΠ. avons constaté qu'il n'y avait pas de système de suivi permettant de τα συστήματα αυτά λοιπόν πρέπει να είναι σε θέση να υποστούν ενδελεχή οικονομικό ε, και λογιστικό έλεγχο με τρόπο ώστε να είμαστε σε θέση να μετρήσουμε την επίπτωση των άμεσων ενισχύσεων μέσω των διαφόρων μορφών αυτών των ενισχύσεων ε, στις κτηνοτροφικές παραγωγές. Κοιτάξτε, δυστυχώ ο εισηγητή σα λόγω οικογενειακών προβλημάτων, από ό,τι μα είπατε, δεν είναι εδώ. Τι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκερμπράντι αλλά και τους συνεργάτες του για το πνεύμα το ανοιχτό πνεύμα και το πνεύμα καλής συνεργασίας το οποίο έδειξε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κρέτα. Έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος ε, επιθυμεί να πάρει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον συγκητή και το Ελεκτικό για το έργο τους και για τις συστάσεις τους. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να κάνω μια διάκριση αυτής εξ αρχής. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του να συζητούμε γενικά για τη συνδεδεμένη υποστήριξη, ενίσχυση και από το να μιλάμε συγκεκριμένα για στήριξη των ε, φυλαζουσών αγελάδων και λοιπόν. Είναι ένας τομέας που με πολλές αναλύσεις είδαμε ότι είναι πιο ευαίσθητος αν δεν υπάρχει στήριξη σε συγκεκριμένες περιφέρειες και είναι δύο είδη περιφέρειων και δύο είδη κινδύνων. Πρώτον, όταν θα είχε η έλλειψη στήριξης περιβαλλοντικό, αρνητικό βέβαια αντίκτυπο, έτσι είναι η γενική εκτίμηση του κινδύνου από όλου ε, τους περιβαλλοντικούς οργανισμούς, ομάδε κτλ. Και, και το έχουμε συζητήσει στα πλαίσια της αναλύτης αντικτύπου. Υπάρχει και υπάρχουν και άλλοι τομεί όπου είναι οικονομικό ο κίνδυνο, οι περιοχέ δηλαδή. Αν δεν υπάρχει στήριξη, παραγωγή, θα στραφούν σε πιο κερδοφόρα είδη παραγωγή. Με μείζωνα πλέον κίνδυνο η... τα αγροτεμάχια να μετατραπούν μόνιμα σε κάτι άλλο. Και αυτό είναι πρόβλημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στόχευση και τι συστάσει σχετικέ, συμφωνούμε με το Ελληνικό συνέδριο ότι η καλύτερη στόχευση πρέπει να είναι ένα από του βασικού ε, προσανατολισμού τη μεταρρύθμισης τη ΣΚΑΠ και το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν και συγκεκριμένα άρθρα τη πρότασή μα προ αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, πρέπει επίση να λάβουμε υπόψη στο το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά, πάντοτε αυτά που σε τέτοιες περιπτώσεις ε, έχουν τη μεγάλη σημασία λόγω των ιδιαιτεροτήτων της δημορφίας. Έχετε και κάποια γραφήματα. Στο πρώτο γράφημα της έκτασης ε, του Ελεκτικού Συνέδρα 19 βλέπετε μια τελείως διαφορετική εξέλιξη ε, του ζωικού κεφαλού δηλαδή να αγελάδων στην Γαλλία και στην ε, Γερμανία. Είναι η ε, που στην Γαλλία κυρίως χρησιμοποιείται η υπαγωγή βοή κρέατος, ενώ στη Γερμανία το αντίστοιχο σωστό είναι 14% εφόσον από τις γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες ε, γίνεται, η... έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής βόη Άρα έχουμε διαφορές στα κράτη-μέλη. Και πρέπει αυτά να μπορούν να αποφασίζουν τι θα κάνουν. Έχοντας βέβαια υπόψη κάποια κριτήρια που πρέπει να παρακολουθεί η Κομισιόν. Και συμφωνούμε απόλυτα με την παρατήρηση αυτή του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτό εξηγεί τα πρώτα δύο σημεία που ανέφερε στην παρέμβαση του κ. Κρετά. Το τρίτο που θέλω να τονίσω είναι ότι η πρότασή μας ε, για τη μετακίνηση της ΚΑΠ περιλαμβάνει και μέχρι τώρα στις διαπραγματεύσεις δεν αμφισβητήθηκε ένα σύστημα παρακολούθησης ελέγχου που θα καλύπτει το σύνολο της κοινή γεωργικής πολιτικής, όχι τα μεμονωμένα στοιχεία. Με τη λογική της δημόσιας παρέμβασης ε, συντατικοποίησης και θα παρέχει και μια σειρά δικτών για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της πολιτικής και να δούμε πού πρέπει να γίνουν αλλαγές. Εδώ ολοκληρώνω και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννίτη. Στις 6.30 πρέπει να πάμε στην Προεδρία της Λιθουανίας. Μπορούμε, έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Θα τα εξαντλήσουμε. Κύριο Ντί, να συγχαρώ τον κύριο Κρετά για την εξαιρετική του έκθεση. Κύριε Πρόεδρε, και αυτό το λέω γιατί με έχει προειδοποιήσει ο Μισελ Ντοντά και το ανακοινώνει εξάλλου και σε άλλες επιτροπές. Αναφέρομαι στις νομοθετικές διατάξεις για να γίνουν σεβαστοί οι στόχοι μας όσον αφορά συγκεκριμένες περιοχές και την τήρηση των στόχων παραγωγής. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί από τη στιγμή που θα συνομοθετήσουμε όσον αφορά τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει σαν αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχής να συνεχίσουμε αυτές τις κατεξουσιοδότηση πράξεις καθότι η πολιτική παρακολούθηση όλων αυτών των πράξεων δεν θα μπορεί να γίνει. Πρόεδρος, ποιος άλλος να πάρει το λόγο. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Κατάλαβα καλά αυτό που είπατε. Ο τριμερής διάλογος είπατε ότι μπορεί να συνεχιστεί με την υπάρχουσα μορφή και μετά το 2013 δηλαδή, χωρίς να αλλάξει. Ποιος μπορεί να απαντήσει η Επιτροπή πρώτα και μετά το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν νομίζω ότι στην παρούσα μορφή του τριμερούς διαλόγου μπορούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε υπόθεση για το ποια μορφή θα πάρει η διαδικασία. Εμείς θα πρέπει να βασιστούμε στα ποσοστά αυτής της στήριξης, της της ε, συνδεδεμένης στήριξης. Τα κριτήρια είναι σαφή. Τα κράτη-μέλη που ζητούν κάτι τέτοιο θα πρέπει να το δικαιολογήσουν. Και βάσει ποιων τομέων ζητούν αυτές τις συνδεδεμένες επιδοτήσεις και στήριξη. Τώρα όσον αφορά τις αλλαγές για τα ποσοστά σε κάποιους τομείς, αυτό ενδεχομένως θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα είμαι όμως εγώ αρμόδιος για αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Κχαϊτά, Πολύ σύντομα. Στη νέα ΚΑΠ ο αριθμός των τομέων που θα μπορέσουν να ζητήσουν αυτές τις συνδεδεμένες επιδοτήσεις, βοήθειες, θα διπλασιαστεί. Κάθε φορά όμως που θα θέλουμε να διατηρήσουμε αυτές τις ε, επιδοτήσεις θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση. Συνεχίζεται δηλαδή κάτι που υπάρχει, συνδυασμός δηλαδή επιδοτήσεων, αλλά με όρους πιο αυστηρούς. Τα κράτη-μέλη δηλαδή καλούνται να δικαιολογήσουν, να τεκμηριώσουν την ανάγκη ύπαρξης αυτών των συνδεδεμένων ε, υποστηρίξεων. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και το Ελεκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή. Χάρη σε εσάς μπορέσαμε να επεξεργαστούμε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ τους συνεργάτες της Επιτροπής, τη Γραμματεία, τα μέλη της Επιτροπής και ευχαριστώ όλους τέλος της συνεδρίασης.

Ευχαριστώ